Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à... Καλημέρα σας. Σας εύχομαι καλώς ήρθατε σε μια σημαντική ψηφοφορία μετά από μια πολύ σημαντική επίσης ε, συμβαστική προσπάθεια που έγινε και θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την εισηγήτριά μας την Μπάρπαρα αλλά και το Συμβούλιο, το οποίο τη γνώμη θα ακούσουμε εντός ολίγου. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την οδηγία που αφορά την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών σε εμπορικέ συναλλαγέ. Μετά από διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο στα πλαίσια του άτυπου τριμερού διαλόγου ε, στην πρώτη ανάγνωση, Φτάσαμε σε αίσιο πέρας και θα δώσω το λόγο στην πρωταγωνίστρια αυτής της επιτυχίας, την Μπάρμπαρα Βάιλερ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα καταλαβαίνετε ότι με κάποια ικανοποίηση, με κάποια περηφάνεια θα σας παρουσιάσω το αποτέλεσμα που λάβατε χθες το βράδυ. Από το αποτέλεσμα και μόνο αντιλαμβάνεται κανείς ότι με το νομοθέτημα αυτό καταβάλαμε προσπάθειες να πετύχουμε το στόχο της καλύτερης νομοθεσίας. Δεν είναι πολύ απλό το νομοθέτημα αυτό, είναι όμως πιο απλό από πολλά άλλα που ε, υιοθετούμε εδώ. Χαίρομαι που πετύχαμε τόση μεγάλη συνένεση. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον σκληρό πυρήνα της ομάδας που μαζί μου και σε συνεργασία με την Κομισιόν και το Συμβούλιο και την, ε, και την Επιτροπή προετοίμασαν το, ε, την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ τον κύριο Χάνσλι Κρότσμαν, ε, Ρούλε, τον Ιόγκ και Κοσνίτσκι. Πιστεύω ότι ο νόμος αυτός όταν θα εφαρμοστεί θα εισάγει μια νέα νοοτροπία ε, στην Ευρώπη, κάτι που θα επωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο νόμος αυτός αποτελεί αποτέλεσμα της ε, πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι έχουμε εδώ μια οδηγία χρήσιμη σε αντίθεση με την προηγούμενη. Τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια θα δούμε βελτιωμένη ρευστότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπω ήδη ότι ως αποτέλεσμα της συζήτησής μας κάποιοι εθνικοί νόμοι διαμορφώνονται και υιοθετούνται. Οι κάτω χώρε, ε, η Βρετανία, ε, η Γαλλία το έχουν ήδη. Στην Ισπανία ετοιμάζεται κάτι αυτή τη στιγμή, ώστε να δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η δυνατότητα μέσω καλύτερη ρευστότητας ε, να επενδύουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ε, νέα προϊόντα. Μία επίκριση θα ήθελα να θυμίσω όλους εδώ στην αίθουσα ότι πρόκειται περί συμβιβασμού. Εάν μπορούσε να αποφασίσει το ε, Κοινοβούλιο μόνο του θα είχαμε 9% τόκο υπερημερίας, δεν θα είχαμε τόσες εξαιρέσεις και θα είχαμε πιο αυστηρή νομοθεσία. Έχουμε όμως 27 κράτη-μέλη και για κάποιο από αυτά οι αυστηροί μας κανόνες ήταν υπερβολικοί και δεν ήθελαν να στηρίξουν την, ε, την νομοθετική αυτή πράξη και τα 27 κράτη-μέλη είναι ε, συνομοθέτης. εξετάστηκαν όλες οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου, δεν υπήρξαν δυσκολίες. Υπάρχουν ε, όμως ε, κάποιοι που τώρα που αποφασίστηκαν όλα στην ε, Κορεπέρ, στο, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, συνεχίζουν να αμφισβητούν το αποτέλεσμα με άσχημες εκστρατείε. Θα ήθελα λοιπόν να το επικρίνω αυτό και ελπίζω σε δύο εβδομάδες να εγκριθεί στην Ολομέλεια η νομοθετική αυτή πράξη που βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον τρόπο που έχουν ετοιμάσει η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Θα δώσω εντάχει το λόγο στους και οδησηγητές. Πρώτα στην κυρία Μαγκοζάτα Χάνσλικ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τη Μπάρμπαρα αλλά και τους υπόλοιπους και οδησηγητές γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετική η συνεργασία μεταξύ μας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά και χάρη στις προσπάθειες και της εισηγήτριας αλλά και των σκιωδών εισηγητών καταφέραμε να καταλήξουμε σε αίσιο πέρας. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω αυτό που είπε η Μπάρβαρα, ότι πρόκειται για συμβιβαστική λύση. 27 χώρες και έχουμε και 27 διαφορετικές γνώμες. Αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι παρά τις διστάμενε διστάμενες απόψεις κατορθώνει και καταλήγει στις συμβαστικές λύσεις. Και αυτό το έγγραφο είναι καρπός μιας τέτοιας συμβαστικής λύσης. Χάρη στην πρόταση αυτή θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανακτήσουν εγκαίρως και εμπρόθεσμα τις ελιξιπρόθεσμες τους ε, αξιώσεις και, ε, ή να πληρώσουν ε, κάπως καθυστερημένα και να μην χρειάζεται λόγω αυτής της καθυστέρησης να οδηγηθούν στην πτώχευση και να πρέπει να εκαθαρίσουν τις επιχειρήσεις τους. Μην ξεχνάτε ότι διανύουμε μια οικονομική κρίση και πιστεύω ότι χάρη στην πρόταση αυτή θα διευκολυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση και η καθημερινή του λειτουργία. Ευελπιστώ ότι θα υποστηρίξετε όλοι αυτό το έγγραφο και σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για τη συνεργασία. Ε, ο κύριος Κρότσμαν απουσιάζει. Κυρία Ρούλε, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και εγώ τους κοιόδης και την εισηγήτρια. Να ευχαριστήσω και την Βελγική Προεδρία, όχι όμως το Συμβούλιο. Χωρί το Συμβούλιο θα ήταν πολύ καλύτερη η νομοθετική αυτή πράξη. Η Βελγική Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά ήταν δύσκολη η κατάσταση εκεί. Η καλύτερη νομοθεσία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μάθει και ο άλλος συνομοθέτης. Cela a le mérite d'être Εντάξει. Ούτε ο κύριο Κωσούσνικ ε, είναι παρόν. Κύριε Ντεγιόγκ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, είναι μια πολύ αξιόλογη επιτροπή. Το θέμα αυτό ήταν ε, από τα πιο ενδιαφέροντα, το θέμα των υπερήμερων πληρωμών και είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα γιατί είναι ένα συγκεκριμένο πολύ απτό θέμα που αφορά το, τους πολίτες. Και χαίρομαι για τις εξελίξεις γιατί παρά την ε, αρχική αντιπαράθεση κατορθώσαμε τελικά να καταλήξουμε συμβαστικές προτάσεις και νομίζω ότι βοήθησε αρκετά η Βελική Προεδρία σε αυτό. Μπορούμε κάλλιστα να υποστηρίξουμε το κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί και ελπίζω ότι θα το κάνουμε. Άλλος κανείς, πέραν του σχεδόν εισηγητών, πως θέλει το λόγο πριν την ψηφοφορία. Αλλιώ να δώσω το λόγο στην Βελική Προεδρία, στον κύριο Βανάμπελε γιατί μετά από τις προσπάθειές σας σας αξίζει να σας δώσουμε το λόγο έστω και για ένα δίλεπτο. Euh, Ευχαριστώ, Προέδρε. Εξ ονόματο Βελική Προεδρία και τη Αντιπροσωπεία μου, θα ήθελα με τη σειρά μου να σα ευχαριστήσω και προφανώ ε, την εισηγήτριά μα, την κυρία Σλίκ, τον κύριο Μπαλταζάρη, τον κύριο Κρέτσμαν, Χουίλε, ε, Ντε Γιούγκ. Ε, προφανώ και τον κύριο Χάρμπορ, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ε, που είχε καταλητικό ρόλο ε, κάποιες στιγμές. Επίσης, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία των Θεσμικών Οργάνων αλλά και τη Νομική Υπηρεσία που πραγματικά κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες. Όλοι οι συνάδελφοι, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μην το ξεχνάμε, ε, επιτέλεσε σημαντικό έργο ούτως ώστε να βρούμε μια κοινή κατεύθυνση. Τώρα, ε, είναι η καλύτερη δυνατή συμβαστική λύση που μπορεί κάποιος να φανταστεί, όχι, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή συμβαστική λύση ε, και είναι ωραίο το αποτέλεσμα και μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. Λοιπόν, πρόκειται για οδηγία ελάχιστη εναρμόνιση και θα απαντήσω στην κυρία Βάιλερ που λυπάται για το 8% μα είναι το ελάχιστο όριο. Οποιοδήποτε κράτος μέλος το επιθυμεί μπορεί να υπερβεί ε, το ελάχιστο αυτό όριο του 8% σε αυτήν την ε, οδηγία ε, και αποδίδω όλα τα εύσημα στο Κοινοβούλιο διότι εγγράψατε σταθερές αρχές και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στην οδηγία και εδώ είναι η πινελιά του Συμβουλίου με κάποια ευελιξία σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του κειμένου. Όπως ακούσαμε και από κάποιους σκιώδεις, ε, ε, θα πρέπει τώρα να ε, σηκώσουμε τα μανίκια, να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η οδηγία. Συγχαίρω όλους όσους εργάστηκαν για αυτό το νομοθέτημα. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ευελική Προεδρία. Ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με μια τέτοια οδηγία. Η Μπάρμπαρα το τόνισε πόσο δύσκολο ήταν να καταλήξουμε συμβαστική λύση. Έχουμε τρία θεσμικά όργανα. Όταν έχουμε μια ευφυή συνεργασία ανάμεσά του, έχουμε και ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ε, η κυρία Μπρίκμαν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο, γιατί και η Επιτροπή κατέβαλε πάρα πολύ μεγάλε προσπάθειε. Ε, ευχαριστώ, πρόεδρο. Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Ευχαριστώ την κυρία Βάιλερ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε με τη βοήθεια όλων των σχεδόν εισηγητών. Ε, από κοινού ε, καταλήξαμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Ήταν δυσχερείς οι εργασίες μας, ε, διότι είναι αρκετά φιλόδοξη αυτή η οδηγία ε, και έχουμε ικανοποιηθεί από το τελικό ε, κείμενο, από το τελικό συμβαστικό κείμενο, διότι παραμένει φιλόδοξη η συμβαστική αυτή λύση. Ε, είναι πιο ευέλικτο το κείμενο, προσθέτει, έχει προστιθέμενη αξία και ο κλάδος, οι επιχειρήσεις αλλά και η αγορά εργασίας ανέμεναν με μεγάλη ανυπομονησία αυτή την ε, οδηγία και νομίζω πως ε, μπορούμε να ελπίζουμε ε, ότι ταχύτατα θα εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα και θα προσφέρει πολύτιμη αρρωγή στις εταιρείε, κυρίως δε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Ωραία, ας περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. 16 από το ΕΛΚΑ. Έχουμε δύο υπεράριθμοι. Έχουν όλη την κάρτα, την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας, παρακαλώ. Καλώς, θα... για να μετράμε είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. c'est pareil. Je vais faire un essai. Je vais faire un vote PPE comme le président. Oui, alors on va faire simplement un vote PPE. Θα κάνουμε μια ψηφοφορία ΕΛΚ για να εξακριβώσουμε τι έχει γίνει. Μόνο ε, το ΕΛΚ ε, ψηφίζει για να μετρήσουμε. 14, c'est bon. 14. Ωραία. Α, 15, 16. Ναι, όντως, ε, δύο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Non, il y a deux Τρεις παραπάνω είναι, 17. Ε, μπορείτε να συνεννοηθείτε παρακαλώ. Il Κάποιοι μαθητές είναι αφηρημένοι σήμερα. Πειράζει. Συγγνώμη, μπορείτε να το ξανακάνετε. Κατά λάθο ε, ψήφισαν ω ΕΛΚ δύο πράσινοι. Et euh, les mêmes voteront, hein Il en manque deux. Ah, un Il en manque un. Ένας ε, επιπλέον. Οι ίδιοι παρακαλώ να ψηφίσουν και στην ψηφοφορία για να μην έχουμε παραπάνω μέλη. Ψηφίζουμε. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστικής πρόταση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Η δική μου κάρτα δυστυχώ δεν λειτουργεί. voilà, c'est bon. 29 euh, ψήφισαν. Παμψηφί υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα η πρόταση. Συγχαρητήρια θερμά κύριε Συγγήτρια. Ah, Ο κύριο Τενταφυλλίδης. Ξέχασα την κάρτα μου, αλλά ψήφισε υπέρ. Ψηφίζω υπέρ. Μπορείτε να συνυπολογίσετε και τη δική μου ψήφο δηλαδή. Zero Χωρίς αποχές, καμία δική ψήφο. Συγχαρητήρια θερμά σε όλους συνεργάστηκαν για το θέμα αυτό. Θα δώσω τώρα και το λόγο και την Προεδρία στην Κάρεν Στήλερ, γιατί θα περάσουμε σε τελείως διαφορετικό θέμα. Η Κάρεν Στήλερ θα μας μιλήσει για τα υλικά δόμησης.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 Ήθελα να ε, ησυχάσετε παρακαλώ. Όσοι θέλουν να μείνουν ε, μπορούν να μείνουν, όσοι θέλουν να φύγουν ε, να φύγουν. περνάμε τώρα στα δομικά προϊόντα. ήδη έχουμε καθυστερήσει λίγο και έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές μαζί μας εδώ σήμερα. Θα θέλαμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όσους σκοπεύετε να παραμείνετε και οι σκιώδεις εισηγητές είναι εδώ και προχωράμε στην ακρόασή μας. Το πρώτο μέρος της ακρόασης έχει να κάνει με την υπερσήμανση CE και τον κανονισμό για τη διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων. Και εξετάζουμε τις βασικές πληροφορίες ε, για την επισήμανση CE για τα δομικά προϊόντα και σε σχέση με άλλα προϊόντα, ποιες είναι οι διαφορές και όχι, τι θα πρέπει να αναφέρεται και τι όχι όσον αφορά την δήλωση απόδοσης, ε, τι γίνεται με τις επικίνδυνες ουσίες και τι σημαίνει σημαίνει στην πράξη όλα αυτά, Ποιε ε, είναι οι συνέπειε ε, των αποκλήσεων που πρότεινε το Συμβούλιο στην ε, θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση στο άρθρο 5 και έχουμε να εξετάσουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την δήλωση απόδοση. Βρισκόμαστε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι τη συζήτησή μα και έχουμε τρει εξαιρετικού ομιλητέ, τον κύριο Γκρέκ Κούπερ που είναι πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνική Έγκριση ΕΟΤΑ, τον κύριο Τζαν Κάρλο Μπετότη, για τα δομικά προϊόντα σύμβουλο και τον κύριο Βινσέντε Λέο Αργέλες ε, που είναι ε, τμήματάρχη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τον γνωρίζουμε πολύ από εμά. Να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Κούπερ να ακούσουμε την παρουσίασή του. Ευχαριστώ. Ε, ναι, φαίνεται να λειτουργεί και η τεχνολογία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Όπως είπε η Πρόεδρος, λέγομαι Greg Cooper. Ε, είμαι ε, διευθυντή στο BBA στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι ένας ε, φορέας έγκρισης. Σήμερα όμως μιλώ εκ μέρους της ΕΟΤΑ. Θα σα παρουσιάσω σήμερα πολύ σύντομα τρία βασικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το CPR, τα, οποία, ε, τα περισσότερα από τα οποία έχουν να κάνουν ε, με τις ε, αρμοδιότητες που αναθέτει σε άλλους η Κομισιόν. Να σας μιλήσω λίγο για τον ΕΟΤΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης. Έχουμε 45 μέλη. Ε, πολλά από τα μέλη είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε ένα μείγμα δημοσίων και ιδιωτικών ε, φορέων. Η ΕΟΤΑ έχει δύο ε, υπαλλήλου εδώ στις Βρυξέλλες. Κατά τα άλλα, μας υποστηρίζουν μέλη με εθελοντική εργασία, όπως κάνω εγώ άλλωστε. Έχουμε εκδίδουμε περίπου 2.000 ε, εγκρίσεις για τις τεχνικές προδιαγραφέ το χρόνο. Και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέλουμε να ενθαρρύνουμε το εμπόριο και ε, την έγκριση νέων δομικών προϊόντων και το 63% περίπου των αξιολογήσεών μας έχουν γίνει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλήσαμε με τους ε, ανθρώπους που λαμβάνουν τις τεχνικές αξιολογήσεις ε, και το βασικό έβριμα μας είναι ότι τους ενδιαφέρει η ε, διαδικασία και τους ανησυχεί κυρίως ο χρόνος. Ο χρόνος είναι πιο σημαντικός από το κόστος, διότι ε, όταν μιλάμε για τις ε, επενδύσεις τους και αυτά, ο χρόνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τους ενδιαφέρει το περιεχόμενο και η συνέπεια των τεχνικών αξιολογήσεων. Οι χρήστες το, της επισήμανσης CE θα πρέπει να γνωρίζουν τι σημαίνει η επισήμανση αυτή. Ένα από τα θέματά μας είναι εάν ε, οι τεχνικές ε, απαιτήσεις αυτές ε, θα οδηγούσαν σε ε, καινοτομία, διότι το να καινοτομεί κανείς, να επενδύει και να μην κερδίζει από αυτό, αυτό δεν είναι καλό. Όπου υπάρχει HEN αλλά δεν είναι χρήσιμη η η μέθοδος ή δεν υπάρχει τέτοια μέθοδος ή έχουμε τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τέτοιο HCN, e οπότε ε, η καινοτομία μπορεί να είναι περιορισμένη ή να έχουμε νέα χρήση ε, μιας εφαρμογής. Ε, με το UNIS υπάρχει ε, κίνδυνος ε, να υπάρχει σοβαρό ε, κενό για τους ε, χρήστες, σοβαρό κενό γνώσης. Προσπαθούμε λοιπόν να το συμπληρώσουμε αυτό για να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση των καινοτόμων προϊόντων. Πιστεύουμε ότι οι διανομής δομικών προϊόντων προσπαθούν να επηρεάσουν τους χρήστες να υιοθετήσουν, να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα προϊόντα. Και προσπαθούν να μεταφέρουν πληροφορίες στους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτού που λαμβάνουν ε, τέτοιες αποφάσεις είναι, ανήκουν ήδη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσο αυξάνεται η καινοτομία θα Αυτό θα είναι θετικό. Μπορεί όμως ε, να υπάρχει σε μεγάλες ε, επιχειρήσεις η εσωτερική επιρογνωμοσύνη για να ερμηνεύονται τα νέα ε, δεδομένα που λαμβάνονται και στον τομέα των οικοδομών αυτή τη στιγμή όσον αφορά την καινοτομία Ε, γενικά αυτές υπόκεινται σε εθνική έγκριση. Επίσης έχουμε τις ε, ευρωπαϊκές ε, τεχνικές αξιολογήσεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προσπαθούν να αντιγράψουν τις εθνικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα θέματα που συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο ορισμός, το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών τεχνολογικών τεχνικών αξιολογήσεων. Ε, έχουμε συζητήσει πολύ τις ε, ευρωπαϊκές ε, τεχνολογικές αξιολογήσεις. Μας απασχολεί ότι για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ειδική. Ε, φοβόμαστε ότι αν διαρκεί πολύ η διαδικασία, τόσο πιο ακριβή θα γίνεται επίσης. Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το EAD και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή του, προϊόντος του προϊόντος κατάλογο των τεχνικών χαρακτηριστικών. Θα πρέπει να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές που, είναι, ε, που ενδιαφέρουν το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να ε, συνδυάζεται με ε, τις τεχνικές προδιαγραφές. Αυτά όσον αφορά το περιεχόμενο και όπως σας είπα συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό. Προφανώς ένα σημαντικό θέμα είναι να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του οικονομικού μοντέλου για όλους όσους συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και τους παραγωγούς αλλά και τις, τους φορείς έγκρισης και ο σχετικός κανονισμός το λαμβάνει αυτό υπόψη στον, ε, στο άρθρο 20 ε, και στο άρθρο 32. Ε, το άρθρο 20 λέει ότι ο καινοτόμος κατασκευαστής δεν θα πρέπει να φέρει μόνος του το κόστος για την έγκριση. Αυτό είναι πολύ λογικό, αλλά ποιο θα είναι το οικονομικό μοντέλο για ε, το EAD. Το άρθρο 32 αναφέρει κάποιους τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό, αλλά όπως πάντα ο διάβολος ε, βρίσκεται στη λεπτομέρεια και συζητάμε με την Κομισιόν τον τρόπο χρηματοδότησης. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει πού δαπανώνται ε, πού προκύπτουν ε, οι διάφορες δαπάνες. Εάν χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα EAD, πόσο στοιχίζει αυτό, ότι γίνεται με την ε, τεχνική αξιολόγηση όταν, για να εκπονηθεί αυτή και δείχνει και το κόστος της, ε, της δαπάνης, λέει, της γραμματείας της ΕΟΤΑ. Αυτά τελικά Το πώς αυτά χρηματοδοτούνται είναι... μια, είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Όσον αφορά λοιπόν ε, το EAD, το European Assessment Document, ε, αυτό το συζητάμε ακόμα με την Κομισιόν. Τα βασικά σημεία λοιπόν για το οικονομικό μοντέλο είναι τα εξή. Ε, πολλοί από τους φορείς ε, όταν αυτοχρηματοδοτούνται ή κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, ο κανονισμός άλλωστε ενθαρρύνει τους φορείς να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και τι γίνεται με το κόστος του EAD, του Ευρωπαϊκού Εγγράφου Αξιολόγησης. Για να εφαρμοστεί ο κανονισμός χρειάζεται ένα καλό οικονομικό μοντέλο, αλλά οι λεπτομέρειες θα πρέπει να εκπονηθούν. Τέλος, όσον αφορά την ε, πρακτική διαδικασία, προσπαθούμε να κινηθούμε εδώ σε θέματα εφαρμογής του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα. Όσον αφορά τα γενικά άρθρα, ο ε, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με τον κανονισμό και τις προτινόμενες τροπολογίες. Αυτό που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή δεν είναι τα απαραίτητα άρθρα, αλλά μάλλον τα παραρτήματα. Το παράρτημα 2 εξετάζει την διαδικασία για την εκπόνηση ενός EAD και έχουμε ανησυχίες ότι ε, γίνεται προσπάθεια να υπάρχει μια διαδικασία η οποία να εφαρμόζεται σε όλους για να οι τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή να καλύπτουν ε, τα πάντα από μια μικρή παραλλαγή ενός προϊόντος ε, που ήδη καλύπτεται από κάποιο πρότυπο μέχρι κάποιο καινοτόμο προϊόν το οποίο δεν έχει δει κανείς ποτέ στην αγορά. Ένα παράδειγμα είναι ότι ζητάει από τον ε, πράκτορα και τον κατασκευαστή πολύ νωρίς να κάνουν ε, αξιολόγηση και όταν μιλάμε για καινοτόμα τεχνολογία ε, μιλάμε για το στάδιο πριν την αξιολόγηση. Αυτό νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει το να εκπονηθεί δηλαδή μια χρήσιμη σύμβαση τη στιγμή που δεν γνωρίζει Κανεί τι είναι το προϊόν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε θέματα πολιτικής. Μου φαίνεται ότι μπαίνουμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες όσον αφορά τι χρονικέ προθεσμίε. Λέει για παράδειγμα ότι η ανωτέρω σύμβαση ε, θα πρέπει να συνάπτεται εντός ενός μηνός ε, σε μια διαδικασία που θα διαρκέσει μάλλον 18 μήνες μέχρι να, ε, να εκδοθεί ε, το, η τεχνική αξιολόγηση. Είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία αυτή. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί το, αν θα πρέπει να είναι ένας μήνας ή έξι, μήνες, ε, ή, έξι εβδομάδες ε, δεν μας φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικότερο, ε, σημαντικότερο είναι ο βασικός μας στόχος. Η θέση μας λοιπόν είναι ότι η λεπτομερής διαδικασία θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους ενδιαφερομένους σε, μια διαφανή διαδικασία. Μπορούμε να πετύχουμε περισσότερη διαφάνεια αν συνομιλούμε με διάφορες ομάδες ε, ενδιαφερομένων. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνεται κατανοητή η διαδικασία. Όπως ε, σας είπα, ε, το έχουμε ξαναθίξει αυτό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπετε εδώ μία μικρή διαφάνεια, μια διαφάνεια που έχει να κάνει με την διαδικασία Βλέπετε εδώ τον ε, κύκλο ζωής και το και θα πρέπει να Η πείρα μας μας δείχνει ότι με καινοτόμα προϊόντα έχουμε ένα αρχικό προϊόν το οποίο θέλουμε να εγκριθεί και να αναπτυχθεί η τεχνική αξιολόγηση με βάση αυτό. Η πείρα μας δείχνει ότι μετά έχουμε ένα δεύτερο ή τρίτο προϊόν που τα οποία μπορεί να διαφέρουν ελαφρά ή να έχουν κάπως διαφορετική χρήση ή άλλες εφαρμογές. Εμείς λοιπόν θέλουμε το EAD, το ε, έγγραφο αξιολόγησης, να να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε τελικά να έχουμε τρία διαφορετικά προϊόντα με τρία διαφορετικά EADs. Τελικά να καταλήγουμε σε μια ομάδα προϊόντων βάσει τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση. Και πιστεύουμε ότι αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν τελικά σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Πιστεύουμε ότι αυτό γίνεται τελικά και θα θέλαμε αυτά να αντικατοπτρίζονται στην ε, συμφωνημένη διαδικασία. Στην επόμενη μου διαφάνεια. Βλέπετε άλλο ένα παράδειγμα παρατήματος ε, το οποίο θα πρέπει να επανεξεταστεί. Το παράτημα 4 ε, εξετάζει το πεδίο εφαρμογή των ε, φορέων έγκρισης. Ο πίνακας 1 όμως είναι κατάλογος κατηγοριών προϊόντων που όμως δεν κοιτάει το μέλλον είναι μάλλον οπισθοδρομικός. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς ποια θα είναι τα καινοτόμα προϊόντα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ορίσει κανείς τους τομείς του οποίους θα εμπίπτουν στον πίνακα 1. Πιστεύουμε λοιπόν ότι απαιτείται εδώ περισσότερη σκέψη, διότι υπάρχει ο κίνδυνος σημαντικής καθυστέρησης κατά την προσπάθεια ορισμού προϊόντων που δεν εμπίπτουν ε, ε, με την πρώτη ματιά σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε μία προσέγγιση πιο ευέλικτη η οποία να βασίζεται ε, στις ικανότητες και πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί σημαντική ότι εδώ υπάρχει η δυνατότητα να ε, δημιουργηθεί κάτι καλό ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα πρέπει να δείξουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στους φορείς έγκρισης. Όσον αφορά λοιπόν τη διαδικασία και την πρακτική εφαρμογή, υπάρχει ανάγκη ε, Βελτίωση των παραρτημάτων 2 και 4. Αυτά μπορούν να γίνουν με ε, ε, πράξη κατοξιδότηση. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι ζωντανή και να βελτιώνεται συνεχώς. Πιστεύουμε επίσης ότι πιθανή λύση θα ήταν μια διατομεακή ομάδα ενδιαφερομένων, κάτι που θα συμβάλλει και στην διαφάνεια. Και αυτό θέλουμε να λυθεί τώρα. Δεν περιμένουμε, δεν σκοπεύουμε να περιμένουμε τον κανονισμό ε, πρωτού θίξουμε θέματα διαφάνειας. Φέτος τον Νοέμβριο θα γίνει ένα εργαστήριο στο οποίο θα συμμετέχουν διάφοροι ε, ενδιαφερμένοι για να συζητήσουν το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ε, κύριε Κούπερ, ήταν πραγματικά πολύ κατατοπιστική ανάλυση που μας, έκανε, που μας κάνατε και περιμένουμε με ανυπομονησία το σεμινάριο του Νοεμβρίου γιατί όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για τα θέματα αυτά περιμένουμε με αδημονία και οτιδήποτε τεκμηρίωση έχετε σχετικά. Και αυτό ισχύει και προς όλους τους καλεσμένους μας. Θα ήθελα παρακαλώ να μας δώσετε τα έγγραφα και οτιδήποτε άλλη τεκμηρίωση διαθέτεται. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τζανκάρλο Μπεντότη. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Όταν έλαβα την πρόσκληση για να εκφωνήσω την ομιλία μου και είδα το χρόνο αγόρευσης όλων των ομιλητών, σκέφτηκα, μα συγγνώμη, είναι αδύνατο να είμαι πλήρης για όλα αυτά τα ζητήματα του πρώτου τμήματος στα ακρόασης. Χρειάζομαι περισσότερα από 10 λεπτά. Παρόλα αυτά, θα προσπαθήσω. Θα αρχίσω από το πρώτο ερώτημα, ίσως του προγράμματος της ακρόασης. Γιατί είναι διαφορετικά τα δομικά προϊόντα. Μα γιατί δεν είναι τελικά προϊόντα που είναι έτοιμα προς χρήση από τον τελικό χρήστη, πρόκειται για ενδιάμεσα προϊόντα που έχουν με μόνιμο τρόπο ενσωματωθεί σε ένα δομικό έργο. Οπότε για αυτά τα προϊόντα η αρχή της ασφάλειας εφαρμόζεται μόνο ε, στο βαθμό που αυτά τα δομικά ε, προϊόντα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των επωνομαζόμενων βασικών απαιτήσεων του έργου. Ένα δομικό προϊόν δεν είναι ασφαλές ή μη ασφαλές από μόνο του. Και αυτή η αρχή ε, αυτή η έννοια της ασφάλειας ε, υπερβαίνει ε, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις υλικές του ιδιότητες. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Σχετίζεται με τη χρήση του προϊόντος αυτού στα πλαίσια του συνολικότερου έργου. Και ποιος θα επομιστεί την ευθύνη γι' αυτό. Υπάρχει ένα χάζο αλλά σαφέστατο παράδειγμα αν θέλετε, μια δοκό ε, ε, με, με το μη 30 εκατομμύρια ε, από ξύλο, από ατσάλι, από χάλι, οτιδήποτε. Αν τη βάλετε αυτή τη δοκό πάνω σε δύο τούβλα, σε απόσταση 25 εκατοστών από το πάτωμα και ζητήσω από κάποιον να περπατήσει πάνω στη δοκό, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δυσκολευτείτε. Αν όμως την ίδια δοκό ότι βάλω 20 μέτρα από το έδαφος και σας ζητήσω να επαναλάβετε το πείραμα, κατά πάσα πιθανότητα δεν να το κάνετε, διότι χρειάζεστε κάτι παραπάνω για να νιώσετε ασφαλείς. Ε, ε, θέλετε ε, κάποια προστασία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτηριστικό του προϊόντος. Δεν άλλαξαν όμως οι μηχανικές ιδιότητες της δοκού. Αναλύωτες είναι απλώς. Αλλάζει η χρήση του προϊόντος. Ως εκ τούτου, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας ε, των προϊόντων διαφέρει ε, ε, η σήμανση ΕΚ σε σχέση με άλλες σημάσεις ΕΚ που υπάγονται στις επωνομαζόμενες οδηγίες νέας προσέγγισης. Γιατί δεν μιλάμε για συμμόρφωση με οτιδήποτε, δεν μιλάμε για συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις των έργων ή σε σχέση με κάποιο ευρωπαϊκό πρότυπο. Ε, απλώς, απλώς θα έλεγα πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν έχουν αποκτηθεί με αξιόπιστο τρόπο χρησιμοποιώντας ε, κοινή φρασιολογία, κοινή ορολογία που έχει ε, συσταθεί βάσει του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πιστοποίησης και άρα αυτές οι πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες και ακριβείς. Ένα άλλο σημείο που αναφέρθηκε σε αυτό το τμήμα της ακρόασης είναι η ερώτηση τι πρέπει να δηλώνεται μέσα σε αυτή τη δήλωση απόδοσης. Ε, πόσα ε, χαρακτηριστικά. Ε, η διαδικασία οικοδόμησης καλύπτει πέντε διαφορετικά στάδια ή και περισσότερα. Ε, και παρεμβαίνουν διάφοροι ε, φορείς ε, σε κάθε στάδιο και έχουν διαφορετικές ανάγκες δηλαδή σε σχέση με το τι πρέπει να γνωρίζουν για κάθε προϊόν. Διαφορετικές τεχνικές ανάγκες, διαφορετικές τεχνικές προσδοκίες. Άρα, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατον να καταρτηθεί ε, τέτοιος κατάλογος τεχνικών χαρακτηριστικών. Εξαρτάται από τη θέση στην αγορά του κατασκευαστή. Εξαρτάται ε, από τον τρόπο χρήσης του προϊόντος μέσα σε ένα συνολικό έργο. Ε, ανάλογα λοιπόν με αυτές τις παραμέτρους μπορεί να διαφοροποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του καταλόγου των χαρακτηριστικών. Ε, κατά τη γνώμη μου, επίσης, ε, ε, είναι περίεργο να λέμε, όπως λέμε στο σχέδιο ή σε αυτό που είδα εγώ, ότι για να αποφύγουμε τις κενές δηλώσεις απόδοσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί τουλάχιστον μία απόδοση. Είναι περιττό. Η δήλωση απόδοσης εξορισμού ενέχει ε, αποδόσεις. Αν είναι κενή δεν υφίσταται ε, η δήλωση. Επιπροσθέτως, το να πούμε ότι αν δηλώσετε τουλάχιστον μία απόδοση, τότε παρόλα αυτά θα πρέπει να παριθμίσετε ε, όλα τα χαρακτηριστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά που εμπεριέχει το πρότυπο. Τι σημαίνει να πάγεται αυτό, ότι θα μετατρέψουμε τις δηλώσεις απόδοσης απόδοση σε μια αφηρημένη περιγραφή προτύπων αφενός και αφετέρου ε, η δήλωση ε, ε, θα μετατραπεί σε μία δήλωση των μη δεδηλωθήσεων αποδόσεων. τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Πέραν τούτου, δεν μπορούς, μπόρεσα να βρω καμία απάντηση σχετικά με το ποιος θα πρέπει να καταρτήσει αυτόν τον κατάλογο. Κατά τη γνώμη μου, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες ε, και ασχολούνται με άλλα πράγματα ε, και δεν νομίζω ότι μπορούν να ε, καταρτήσουν ένα τέτοιο κατάλογο, έστω και αν είναι ελάχιστος. Το βασικό χαρακτηριστικό της δήλωσης αυτής, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να είναι ο αριθμός των τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά το ότι η δήλωση απόδοσης ε, εφόσον ε, ε, συνδέεται και με την ανάληψη ευθύνης από τον κατασκευαστή για το τι περιέχεται μέσα σε ένα έργο σημαίνει ότι το προϊόν συνάδει με τα δεδηλωθέντα και ότι η δήλωση έχει εκπονηθεί χρησιμοποιώντας την ε, κοινή ορολογία των ευρωπαϊκών ε, τεχνικών προδιαγραφών. Και πάλι πιστεύω ότι το πεδίο του κανονισμού CPR, όπως λέει ο τίτλος, είναι να δώσει ένα πλαίσιο θέση σε εμπορία. Ε, όχι για τις ίδιες τις αγορές. Τις αγορές, κατά τη γνώμη πρέπει να τις αφήσουμε ελεύθερες να επιλέξουν τι ακριβώς χρειάζονται. και να εκφραστούν δυνάμει του πλαισίου που ε, θεσπίζεται βάσει του σχεδίου κανονισμού. Ε, ένα τελευταίο σημείο θα ήθελα να γύρω που δεν έχω βάλει μες στη διαφάνεια για τις ε, εξαιρέσεις, αποκλήσεις. Ε, αναφέρεται στο σχετικό άρθρο Μάλλον χρησιμοποιούνται τρεις φρασιολογίες. για τους μεμονωμένους πελάτες ε, και τα λοιπά. Σας παραπέμπω στη διατύπωση. Λοιπόν, ε, πόσα κτίρια στις Βρυξέλλες έχετε δει με την ίδια πρόσωψη. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Ε, το κτίριο Μπεγλεμό έχει δική του πρόσωψη. Η Επιτροπή, το κτίριο της Επιτροπής των Περιφερειών άλλη. Ε, πρόκειται για ε, προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί βάσει κάποιων συγκεκριμένων προδιαγραφών προφανώς, αλλά δεν μπορούν να τύχουν ε, εξαίρεσης. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται πολύ καλύτερος ορισμός ε, των μεμονωμένων προϊόντων κατά παραγγελία, custom made, γιατί μετά την έγκριση αυτού του σχεδίου κανονισμού θα προκύψουν διαφορετικές ε, παραπλανητικές ε, ερμηνείες ε, στρεβλώνοντας έτσι την έννοια, το στόχο, τον ίδιο της διάταξης περί εξαιρέσεων. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε, ήσασταν ειλικρινέστατος και το εκτιμούμε. Ας περάσουμε στον τελευταίο μιλήτη ο κύριος Βινσέντο Αργουέλλας, παρακαλώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους σας. Προσπάθησα στην παρουσίασή μου να επικεντρωθώ αυστηρά στα ερωτήματα που θέσατε. Φαντάζομαι είναι τα ίδια ερωτήματα που θέσατε και στους προηγούμενους εμπειρογνώμονες, τον κύριο Μπεντότη για παράδειγμα. Λυπάμαι κύριε Μπεντότη αλλά μερικές φορές είστε καταδικασμένος στο να ακούτε τα ίδια και τα ίδια. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη δυσάρεστο, γιατί ο κύριος Μπεντότη εργάζεται στο ΣΕΝ. Μας βοηθάει λοιπόν στην εκπόνηση των σωστών και χρήσιμων προτύπων. Και είναι λογικό ένας σύμβουλος που εργάζεται στο ΣΕΝ να συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό είπα κύριε Μπεντότη ότι ίσως ε, σας ε, φανούν κάπως ενιαρά αυτά γιατί θα ακούσετε τις ίδιες απαντήσεις στα ίδια ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά καταρχήν τη σήμανση σε Ε για τα προϊόντα δόμησης. Είναι διαφορετική η σήμανση αυτή σε Ε για τα δομικά προϊόντα από ό,τι για τα άλλα προϊόντα. Η απάντηση είναι καταφατική. Είναι διαφορετικό αυτό το σήμα σε για τα προϊόντα δόμησης και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αυτή είναι η πιο σημαντική διαφορά στο όλο εγχείρημα που κάνουμε. Δυστυχώς, πολύ συχνά δεν γίνεται κατανοητή αυτή η διαφορά. Η μέθοδος μου είναι να ακολουθήσω τους ε, ορισμούς ως προς το περιεχόμενο. Τι σημαίνει καταρχήν ε, σήμα σε στις οδηγίες της νέας προσέγγισης. Η επισήμανση σε σημαίνει απλώς συμμόρφωση του προϊόντος με τις ε, βασικές προδιαγραφές ή απαιτήσει ε, ασφάλειας της οδηγίας. Όλοι γνωρίζουμε το πρώτο παράρτημα όλων των οδηγιών της νέας προσέγγισης που αναφέρονται στα ουσιώδη, στις ουσιώδεις απαιτήσει ασφάλειας του προϊόντος του προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας. Για να τεθεί σε εμπορία ένα προϊόν θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες ε, προϋποθέσεις και απαιτήσει. Αυτό εννοούμε όταν εννοούμε συμμόρφωση του προϊόντος με τις ε, βασικές αυτές απαιτήσει. Στην περίπτωση του σήματο Ε για τα προϊόντα δόμηση, δεν μιλούμε ακριβώ για τον ίδιο βαθμό συμμόρφωση. Μιλούμε περισσότερο για απόδοση. Άλλο συμμόρφωση και άλλο απόδοση. Στο παράρτημο 1 του κανονισμού για τα προϊόντα δόμηση, δεν έχουμε πια ε, στοιχειώδεις απαιτήσει για το προϊόν. Γιατί είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε τις στοιχειώδεις απαιτήσει ή προϋποθέσεις για τα δομικά προϊόντα. Το παράρτημα μας όμως μιλά για το πώς λειτουργεί ένα προϊόν. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια γέφυρα για να θεωρείται ασφαλής, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα κτίριο για να θεωρείται ασφαλές. Τι σημαίνει λοιπόν ε, η σήμανση σε ε για τα προϊόντα δόμηση Σημαίνει ότι η δεδηλωμένη επίδοση του απόδοση του προϊόντος έχει ε, ελεγχθεί σε ό,τι αφορά την προτινόμενη χρήση με βάση τα εναρμονισμένα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Εγγράφου Αξιολόγησης. Δηλαδή, σήμα ε, σε ε για τα προϊόντα δόμηση σημαίνει ότι για να είναι αξιόπιστο ένα προϊόν θα πρέπει ο κατασκευαστής να συμμορφωθεί με όλες τις ε, διατυπώσεις, με όλες τις ε, διαδικαστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό. Οπότε, απαντώ στα δύο πρώτα ερωτήματα ότι η δήλωση απόδοσης ε, θα πρέπει να είναι σωστή, ακριβής και ο κατασκευαστής να αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της δήλωσης. Αυτό σημαίνει σήμα σε ε για τα προϊόντα δόμησης, κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από το, από το σήμα σε ε για τα άλλα προϊόντα των οδηγιών νέας προσέγγισης. Άλλωστε στα προϊόντα δόμησης δεν έχουμε καν οριακές τιμές. Δεν προαπαιτείται τίποτα. Και μια και δεν υπάρχουν οριακές τιμές, για τα προϊόντα που τίθεται στην αγορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τα άλλα προϊόντα. Κατ' εξαίρεση μπορούμε να έχουμε οριακέ τιμέ μόνο. Ο κανόνα πάντω ε, προβλέπει ότι στα προϊόντα δόμηση δεν προβλέπονται ή δεν επιβάλλονται οριακέ τιμέ ούτε μέσω των προτύπων ούτε μέσω του κανονισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η απουσία οριακών τιμών. Γιατί λοιπόν έχουμε τόσε πολλέ διαφορέ με τα άλλα προϊόντα. Όπω είπε ο κύριο Μπεντότη, τα προϊόντα δόμησης είναι διάμεσα προϊόντα και από οικονομική και από πρακτική άποψη. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα προϊόντα προκειμένου να ενσωματωθούν σε ένα έργο. Δεν είναι αυθυπόστατα, δηλαδή δεν είναι προϊόντα καταναλωτικά. Φυσικά κατά κάποιο βαθμό μπορεί να έχουν επαφή άμεση με τους καταναλωτές. Πάτε στον πρικό, αγοράζετε τέτοια προϊόντα, έχετε άμεση επαφή κατά, κατά κανόνα. Αλλά αυτό είναι εξαίρεση ακόμη και όταν το αποφασίσει ο ίδιος ο καταναλωτής να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν, δεν είναι καταναλωτής του προϊόντος, δεν το καταναλώνει, απλώς το χρησιμοποιεί. Γιατί αυτό το προϊόν δεν θα το καταναλώσει άμεσα, θα το εντάξει σε μία κατασκευαστική διαδικασία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα προϊόντα δόμησης δεν είναι τελικά προϊόντα, είναι ενδιάμεσα προϊόντα. Και, και η ασφάλεια δεν ισχύει για το ίδιο το προϊόν. Ισχύει για το τελικό αποτέλεσμα, για το έργο. Φυσικά υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές ασφάλεια και για τα προϊόντα. Για παράδειγμα το περιεχόμενο των επικίνδυνων ουσιών. Φυσικά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα προϊόντα δομή θα πρέπει να είναι ασφαλή για τον χρήστη, για τον εργαζόμενο που θα τα χειριστεί. Βάλτε όμως λίγο το μυαλό σου να δουλέψει τι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και πού ρυθμίζονται αυτά. Γιατί αν μιλούμε για ασφάλεια, θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η μόνη εξαίρεση εδώ είναι το περιεχόμενο ή η έκκληση επικίνδυνων ουσιών. Και αυτό ε, προκύπτει από τους κανονισμούς και από του εμπειρογνώμονε που ξέρουν πώ να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Ο συγκεκριμένο όμω κανονισμό προϊόντων δόμηση δεν καθορίζει χαρακτηριστικά ασφάλεια για τα προϊόντα δόμησης. Μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό, αλλά δεν θα βρείτε πουθενά χαρακτηριστικό ασφάλεια. κάτι που να μιλά για την ασφάλεια του προϊόντος δόμησης. Τώρα, υπάρχει μια τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά αυτό το θέμα, το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων δόμησης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, ή μάλλον όχι, βιάζομαι, αυτό είναι για αργότερα το θέμα. Επαναλαμβάνω, η ασφάλεια αφορά τη χρήση του προϊόντος. Πέραν του θέματος των επικίνδυνων ουσιών στο περιεχόμενό του. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να γίνεται σωστή χρήση του προϊόντος δόμησης. Ποιος είναι όμως ο υπεύθυνο για τη χρήση αυτού του δομικού προϊόντος? Ο χρήστης φυσικά. Όπως σε κάθε έκφαση της ζωής, αυτός που είναι υπεύθυνο για το κτίριο δεν είναι ο κατασκευαστής του τσιμέντου, είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο πολιτικός μηχανικός. Αυτή είναι η οργολάβος, αυτή είναι η υπεύθυνη για το κτίριο. Για να μπορούν όμως αυτοί οι άνθρωποι, ο αρχιτέκτονας, ο πολιτικός μηχανικός εργολάβος να, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, χρειάζονται πληροφορίες για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν. Αυτό είναι που χρειάζονται. Και αυτό επεξεργαζόμαστε τώρα, ένα σύστημα ενημέρωσης που θα τη χάνει τέτοια ώστε κάθε παράγοντας της αγοράς, είτε ε, βρίσκεται στην πλευρά της προσφοράς, είτε στην πλευρά της ζήτησης, να καταλαβαίνει από την πληροφορία περί Ποιο προϊόντος πρόκειται. Αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το σύστημα ενημέρωσης και το σύστημα ενημέρωση είναι ουσιαστικά τα πρότυπα και οι προδιαγραφές. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση απόδοσης. Η δήλωση απόδοσης θα πρέπει να αναφέρεται σε μια προτινόμενη χρήση. Λογικό αυτό, γιατί φυσικά ένα προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Πού όμως, πού θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο προϊόν. Οπότε ο αρχιτέκτονας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το προϊόν χρειάζεται πληροφορίες για τη χρήση του. Και τις χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες για πρακτικούς λόγους αφενός και αφετέρου, γιατί μπορεί να ισχύουν κανονισμοί στα κράτη-μέλη που να αφορούν τη χρήση. Δεν έχουμε κανονισμούς ε, γενικούς και αόριστους, αφηρημένους. Έχουμε ένα κανονισμό, για παράδειγμα, που λέει ότι οι μοκέτες στην αίθουσα αυτή θα πρέπει να είναι ανθεκτική στην, στη φωτιά τουλάχιστον 60 λεπτά. Είναι συγκεκριμένοι οι κανονισμοί και αφορούν πάντα τη χρήση του προϊόντος. Κάτι που είναι λογικό γιατί αυτό θα κρίνει στη τελική ανάλυση την ασφάλεια ή την έλλειψη ασφάλειας σε ένα κτίριο. Οπότε τέτοιες πληροφορίες αφορούν κανονικά τη χρήση του προϊόντος. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος καθορίζεται σε σχέση με την χρήση του. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολύ σημαντική έννοια. Εκ των υστέρων γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα ενσωματώθηκαν ε, σε μια διαδικασία γιατί ήταν κατάλληλα για τη χρήση. Και ποιος αποφασίζει αν ένα προϊόν είναι κατάλληλο για μια συγκεκριμένη χρήση? Ο χρήστης, ο αρχιτέκτονας ή ο εργολάβος, όχι ο κατασκευαστής το προϊόντος. Γιατί ο κατασκευαστής θέτει το προϊόν στην αγορά, στην εμπορία, για πολλές χρήσεις. Αλλά εναπόκειται στο χρήστη να επιλέξει την χρήση που θα κάνει. Το Συμβούλιο τώρα αποφάσισε ότι όλοι οι κατασκευαστές που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά θα πρέπει να δηλώνουν τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό που να αφορά την προτινόμενη χρήση. Την χρήση. Ποιο χαρακτηριστικό όμως δεν απάντησε το Συμβούλιο στην ερώτηση αυτή. Κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν απαντά σε αυτή τη σημαντική ερώτηση οφείλεται στο ότι το Συμβούλιο επαφίεται στην αγορά. Το Συμβούλιο είναι βέβαιο ότι η αγορά θα παίξει το ρόλο της και αυτό το πιστεύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι είναι η αγορά. Η αγορά είναι το πρώτο θέτει ε, ένα πλαίσιο ε, προϋποθέσεων τον κανονισμό με, για τη χρήση και μετά γίνεται το παιχνίδι της προσφοράς και της ζήτησης. Υπάρχει το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας με βάση τις προδιαγραφές και τότε ο, κα, κατασκευαστής θα κάνει τη δήλωση ανάλογα με αυτά που απαιτείται από αυτόν. Το Συμβούλιο λοιπόν δεν είναι η απάντηση γιατί θεωρεί ότι η αγορά θα τα ρυθμίσει από μόνη της. Κατά τη γνώμη μας, η λογική του ενός χαρακτηριστικού είναι είτε ότι θα πρέπει να δηλώσετε όλα τα συναφή χαρακτηριστικά για την προτινόμενη χρήση, όπως προκύπτουν στο πρότυπο. Αυτό είναι λογικό, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που είναι συναφή με τη χρήση. Ή μια άλλη λογική που θα μπορούσε να ακολουθήσει το Συμβούλιο ή η Επιτροπή είναι ότι επειδή είμαστε βέβαιοι ότι ο υπεύθυνο χρήστη θα επιλέξει το προϊόν που είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση, δεν χρειάζεται εμείς να, να επιβάλλουμε μάλλον υποχρεώσεις που θα δημιουργήσουν κολλήματα στην αγορά ή άλλα προσκόμματα ή θα επιβαρύνουν με γραφειοκρατία τους κατασκευαστές και τους πολίτες. Αυτές είναι κατά τη γνώμη μας οι μόνες δύο εναλλακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στη λογική. Ή όλα ή τίποτα. Αλλά υπάρχει και ενδιάμεσος τρόπος, ενδιάμεση λύση που είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό. Ούτε όλα τα χαρακτηριστικά, ούτε κανένα. Τώρα, για τις ε, επικίνδυνες ουσίες, θα πρέπει να δηλώνονται ή όχι. Η απάντηση είναι ναι, θα πρέπει να δηλώνονται οι επικίνδυνες ουσίες αλλά υπάρχουν ήδη άλλες νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση δήλωσης τέτοιων επικίνδυνων ουσιών. Και κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει αποχρόν λόγος ώστε αυτή την υποχρέωση να την επιβάλλουμε μόνο στα προϊόντα δόμησης και όχι σε άλλα προϊόντα. Γιατί η νομοθεσία του REACH για τις επικίνδυνες ουσίες ήταν καρπός μιας χρονοβόρας διαδικασίας διαπραγματεύσεων, η οποία έχει καταλήξει σε μια ισορροπία και πρόκειται για μια πολύ δυναμική νομοθετική ρύθμιση. Και όπως λέμε, οι καλοί φράχτες κάνουν τους καλούς γείτονες. Γι' αυτό και καλό θα είναι ο συγκεκριμένος κανονισμός για το προϊόντα δόμησης να μην περιλαμβάνει διατάξεις ε, για τις επικίνδυνες ουσίες, γιατί υπάρχει ειδική ρύθμιση για τις επικίνδυνες ουσίες εκτε, εκτενής που είναι το REACH. Βέβαια, αναφέρθηκε η πρόταση γιατί να μην έχουμε και στον κανονισμό αυτό μια μνήμα που λέει όταν υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις που απαιτούν δήλωση επικίνδυνων ουσιών θα τηρούνται οι αντίστοιχε νομοθετικές διατάξεις και θα ενημερώνονται οι χρήστες για την κατάσταση αυτή. Αυτή, κατά τη γνώμη μας είναι η σωστή λύση. Η μνήμα των αντίστοιχων νομοθετημάτων που προβλέπουν ε, διατάξεις για τη, ή υποχρεώσεις για τις επικίνδυνες ουσίες, αλλά όχι συγκεκριμένες διατάξεις στον κανονισμό αυτό. Για το άρθρο 5. Ρωτήσατε για τις εξαιρέσεις. Είπε και ο κύριος Μπεντότη ότι το 5α Καταρχήν θα πρέπει να προσδιορίζει τι εννοεί εξατομικευμένο προϊόν, θα πρέπει να προσδιορίζει το custom made ή τις διαδικασίες εκτός σειράς. Υπάρχουν αδυναμίες στο άρθρο αυτό κατά τη γνώμη, και, κατά γνώμη μας και καλό θα ήταν να συμπληρωθεί. Το δεύτερο τμήμα της εξαίρεσης με κατέπληξε που το διάβασα γιατί λέει ότι ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια του προϊόντος αλλά φέρει και την ευθύνη αυτών που θα πρέπει να εκτελούν ασφαλώς ε, τα προϊόντα να χρησιμοποιούν ασφαλώς τα προϊόντα αυτά. Τελικά δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Είναι κάπως συγκεχημένη αυτή η εξαίρεση. Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί περαιτέρω. Και κάτι που δεν ε, ρωτήσατε ρητά αλλά επιτρέψτε μου να το αναπτύξω για τις απλουστευμένες διαδικασίες και το STD. Νομίζω ότι έγινε αντιληπτό δηλαδή γιατί προτείνω αυτό το περίεργο ακρονίμιο STD. STD σημαίνει απλώς κατάλληλη τεκμηρίωση. Και αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι ότι όλοι θέλουμε απλουστευμένες διαδικασίες. Θέλουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία και το γραφειοκρατικό άκθος για τις επιχειρήσεις. Όλοι συμφωνούμε ως προς το στόχο αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό τροποποιούμε κάπως τη διατύπωση και λέμε τι μας ενδιαφέρει εδώ πιο πολύ. Μας ενδιαφέρει να προσδιορίσουμε την απλουστευμένη διαδικασία. Και αν θέλουμε απλουστευμένη διαδικασία θα πρέπει να την προσδιορίσουμε σωστά. Και αυτό τώρα γίνεται. Δεύτερο σημαντικό είναι να προσδιορίσουμε πότε, δηλαδή υπό ποιες, προποθέσει μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η απλουστευμένη διαδικασία. Αυτό είναι φυσικά κέριο. Και τέλος θα πρέπει ο κατασκευαστής όταν χρησιμοποιεί την απλουστευμένη διαδικασία να την τεκμηριώνει δεόντως. Οπότε κάθε φορά που βλέπουμε το STD θα πρέπει να καταλαβαίνουμε κατάλληλη τεκμηρίωση ή σωστά τεκμηριωμένο. Αυτό εννοούμε με το STD. Για να αποφευθούν περιτές αντιδικίες και να αποφύγουμε και περιτές και στήρες συζητήσεις. ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις πρώτους ε, ομιλητές. Έχει πάει 4 και 10 η ώρα. Χαίρομαι που έχουμε τον κύριο Ρίπο, την κυρία Αν μαζί μας και άλλους για τη συζήτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν ε, κάτι να πούν οι σκιώδεις. Μία συμπληρωματική ερώτηση όσον αφορά τη δήλωση απόδοσης και τις παρεκκλήσεις. όταν έχουμε παρέκκληση σύμφωνα με το άρθρο 5 και κατά τη δική μου γνώμη δεν είναι διατυπωμένο αυτό πολύ καλά τότε καταλήγουμε σε δυσκολίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 όπου λέει ότι πληροφορίες υπό κάθε μορφή σχετικά με την απόδοση όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά διατίθενται μόνο όταν περιλαμβάνονται και διευκρινίζονται στη δήλωση απόδοσης. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια. Η ερώτησή μου, εάν δεν υπάρχει δήλωση απόδοσης, τότε δεν επιτρέπεται να δίνονται πληροφορίες διότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ε, απόδοση, στη δήλωση απόδοσης επειδή δεν υπάρχουν. Μου φαίνεται ότι εδώ έχουμε ένα μεγάλο κενό διότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να δίδονται πληροφορίες για ειδικά προϊόντα τα οποία έχουν ε, ε, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ε, στα μέτρα του πελάτη. Και μία ακόμα ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Ποια είναι η γνώμη σας, καθώς και των άλλων εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την εξαίρεση, την παρέκκληση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις μικροεπιχειρήσεις. Και όσον αφορά το θέμα της γλώσσας, θα πρέπει ε, τα χαρακτηριστικά απόδοσης να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες. Ε, ένας κατασκευαστής δεν ξέρει ο χοντρέμπορος προς ποιες χώρες πουλάει ε, τα προϊόντα. Θα Πρέπει λοιπόν να παρακολουθεί την πορεία του κάθε προϊόντος του, να ξέρει αν θα κατελήξει στη Γαλλία και να το μεταφράσει στα γαλλικά, αν ε, πωλείται το προϊόν του στην Ελλάδα να ε, δώσει τα στοιχεία στα ελληνικά. Θα ακολουθήσουν και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάιρ. Η Χάιτι Ρίλε. Θα είμαι σύντομη, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πάρουν το λόγο και άλλοι, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς ορίζει η Κομισιόν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όταν ε, στο άρθρο 4 αναφέρεται στα ε, προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται ε, κατά παραγγελία ή προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με αυτό που θέλει ο πελάτης. Και όσον αφορά την επισήμανση λείπει τελείως ε, όρο εποπτεία στην αγορά. Βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία να τα ρυθμίζει όλα η αγορά, αλλά η τιμή παίζει σημαντικό ρόλο και η εποπτεία της αγοράς ε, υπάρχει για να μην ε, αποφασίζονται όλα σύμφωνα με το, την τιμή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό κενό στον κανονισμό ε, περιδομικών προϊόντων το ότι λείπει το τελείως ο όρος εποπτείας αγοράς. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούιλε. Θα παρακαλούσα... Ε, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Α, να ζητήσω από τους ομιλητές μας να απαντήσουν στον κύριο Μάερ και στην κυρία Ρούιλε, αν είναι δυνατόν. Ο κύριος Κούπερ. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Ωραία. όσον αφορά την ε, παραγωγή μικρής κλίμακας και τις παρεκκλήσεις που προβλέπονται. Πιστεύω ότι όλα εξαρτώνται από το πού προέρχεται ο ορισμός του προϊόντος. Τα περισσότερα δομικά υλικά διατίθενται στην αγορά από τους κατασκευαστείς. Η απόφαση σχετικά με την καταλληλότητά τους γίνεται, λαμβάνεται από τον χρήστη. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα τον σχεδιασμό ειδικού παραθύρου για ένα καθεδρικό ναό. Στην περίπτωση αυτή ο σχεδιασμός γίνεται πριν διατεθεί στην αγορά το προϊόν. Υπό τις συνθήκες αυτές, γιατί να είναι απαραίτητο να έχει επισήμανση το προϊόν, διότι εξορισμού τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ε, έχουν ε, τεθεί από τον σχεδιαστή. Αυτές ήταν, ε, αυτή ήταν η συλλογή για το θέμα αυτό. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Κούπερ. Αν κατασκευάζω πόρτες και λάβω παραγγελία να φτιάξω μια πόρτα, να πουλήσω μια πόρτα για τον καθεδρικό του Αγίου, Πέτρου, του Αγίου Παύλου. Ε, δεν θα πρέπει να έχει επισήμανση σε ε, η πόρτα αυτή, διότι είναι κατασκευασμένη ε, κατά παραγγελία, σύμφωνα με συγκεκριμένε προδιαγραφές. Αλλά στο παράδειγμα που σας έδωσα, για παράδειγμα την πρόσωψη του Περλεμό, μπορεί να έχουμε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν σύστημα ενοποιημένου προφίλ, ε, αν θέλετε να παραμείνουμε στο παράδειγμα της συγκεκριμένη πρόσωψης. Ε, και μπορούν, μπορούν ε, οι προδιαγραφές να προέρχονται από μια σειρά άλλων προϊόντων. Αυτά... Αυτά δεν είναι μονομένα προϊόντα επί παραγγελία. Ε, τέτοιο προϊόν είναι η πόρτα του, για το καθαριστικό του Αγίου Παύλου. Η Κομισιόν, ναι, ευχαριστώ πολύ σύντομα, διότι ε, τέθηκαν πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ε, να ξεκινήσω από την τελευταία, τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο το οποίο ε, έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει πολύ ε, καιρός. Ε, λογικά όμως θα πρέπει να υπάρχει ορισμός στην τελευταία εκδοχή του κανονισμού δομικών προϊόντων. Όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης, είναι η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερο, λιγότερους από 10 εργαζομένους. Ε, δύο κριτήρια υπάρχουν, ε, ο αριθμός των απασχολούμενων ε, και το, ο κύκλος εργασιών, ο οποίος δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει νομίζω 250.000 ευρώ. Ο, όσον αφορά τις ε, γλώσσες, ε, σύμφωνα με το άρθρο 37, εάν διαβάσουμε προσεκτικά το άρθρο αυτό, το 37, βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να ισχύει μόνο στις ε, τοπικές επιχειρήσεις. Διότι εκτός από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, άρθρο 37 επαναλαμβάνει ο μιλητής, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικροεπιχειρήσεις. Άρθρο 7-4. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Εντάξει, αυτό προέρχεται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Έχει ήδη γίνει σχετική συζήτηση και λήφθη απόφαση. Έχουμε προσπαθήσει, όπως και το Συμβούλιο, να ακολουθήσουμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό βλέπουμε μπροστά μας. Είμαστε διατεθειμένοι να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό, αλλά έχει αποδειχθεί ότι είναι καλύτερη η ρύθμιση αυτή από αυτό που είχαμε πριν. Όσον αφορά το άρθρο 4.2, πιστεύω ότι... Νομίζω ότι καταλαβαίνω την ερώτησή σας, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι συμμερίζομαι το συλλογισμό σας. Εάν δεν δηλώνεται ένα χαρακτηριστικό, δεν μπορεί να διαφημίσει κανείς το χαρακτηριστικό αυτό. Αυτά με πολύ λίγα λόγια. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε ε, να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσει να δηλώσουν τα χαρακτηριστικά. Εάν δεν το δηλώνετε, δεν το συζητάτε. Νομίζω όμω ότι επί τη αρχή είναι θετική η προσέγγιση αυτή. Ευχαριστώ που απαντήσατε στις ερωτήσεις των ε, συναδέλφων. Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της ε, ακρόασής μας. Ήδη έχουμε καθυστερήσει πέντε λεπτά. Θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το χρόνο. Θα σας ε, παρουσιάσω τους ομιλητές μας. Έχουμε τον Δόκτορα David Μουρ ε, που, είναι, ε, που προέρχεται από την Βρετανία, είναι διευθυντής μηχανικός. Έχουμε τον κύριο Γιάνν Κούμανς που δουλεύει πάνω στις οδηγίες, τα πρότυπα και την διασφάλιση της ποιότητας. Έχουμε τον, κύριο, τον καθηγητή που είναι πρώην ε, πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου για ε, Δομική Τεχνητική ε, Ασχολείται με τους ευρωπαϊκούς κωδικούς. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Και τέλος τον κύριο Μάικλ Ρόμπερτς που εκπροσωπεί την ΚΑΝ, την Επιτροπή για, την εργασία και, για την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας καθώς και για την τυποποίηση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον δόκτωρα David Μουρ Παρακαλώ. Thank you, Chairman. And good afternoon, <clears throat> ladies and gentlemen. Ευχαριστώ. Ε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ σήμερα. Θα σας ε, παρουσιάσω κάποια ζητήματα σχετικά με τη σήμανση ΕΚ ε, για την χαλιβουργία και τις δομικές κατασκευές. I thought I'd perhaps uh, start the presentation. Θα αρχίσω κάνοντας μια επισκόπηση της αγοράς των δομικών υλικών εδώ στην Ευρώπη. Μετά θα μπω σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες ε, για τη χαλιβουργία, ε, για τους κατασκευαστές, μέχρι και την παραγωγή και την ανέγερση. Ο κανονισμός καλύπτει μία πληθώρα δομικών ζητημάτων και πολλά από αυτά τα προϊόντα κατασκευάζονται από τον κλάδο μου. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Ε, το βλέπετε εδώ τη σήμανση και τα, τους διάφορους ε, κλάδους ε. Ε, σας παραπέμπω τώρα στο άρθρο 5 για τις εξαιρέσεις, ε, μετά βιωσιμότητα και αστυνόμευση της σήμανσης. Ε, πώς θα γίνει αυτό. Θα υπάρχουν αρχές επιβολής ε, νόμου ε, ανά την Ευρώπη που θα έχουν τις απαιτούμενε δεξιότητες και αρμοδιότητες για να ε, κάνουν τον έλεγχο, να διεξάγουν τον έλεγχο και με... Λοιπόν, η ο κλάδος εκπροσωπεί 8% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 20 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον κλάδο των δομικών κατασκευών, από τους οποίους έχουμε 8 ε, εκατομμύρια τόνους ε, για διάφορα προϊόντα, από μικρά, ε, από, μέχρι, από δηλαδή, μέχρι σπίτια, αποθήκες, υπεραγορές, ε, ψηλά κτίρια, ουρανοξύστες, ε, γέφυρες, με ευρύτατο φάσμα προϊόντων. Ε, πώς αρχίζει η διαδικασία. Παίρνουμε τον, το μετάλλευμα, το καίμε μέσα ε, ε, στο καμίνι και μετά βλέπετε αριστερά πώς φτιάχνουμε μία τομή και βλέπετε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Ε, δηλαδή, ε, ε, έχουμε χιλιόμετρα τέτοιων χαλίδινων ράβδων που χρησιμοποιούμε και βλέπετε τη σήμανση ΕΚ από τους ίδιους τους κατασκευαστές και οι εργολάβοι αγοράζουν τα χαλιβουργικά προϊόντα και τα επεξεργάζονται ε, ούτως ώστε να φτιάξουν περίπλοκες ε, ε, χαλίβδινες κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια μέσα στα κτίρια. Βλέπετε πώς παρασκευάζονται τα προϊόντα, πώς μεταφέρονται. και ε, τα ίδια τα επεξεργασμένα προϊόντα θα λάβουν μετέπειτα τη σήμανση και θα τεθούν σε εμπορία. Ε, στη συνέχεια φτιάχνουμε δοκούς ε, και άλλα όρθια προϊόντα. Βλέπετε στις τρεις φωτογραφίες που σας δείχνω διάφορους συνδυασμούς προϊόντων, συνδυασμούς ράβδων που χρησιμοποιούνται στο χαλίβδινο πλαίσιο του κτηρίου. Ε, τα προϊόντα που ανήκουν σε ένα συνδυασμό φέρουν σήμανση. Δηλαδή το ή κρύωμα ή οποιαδήποτε άλλη ε, κατασκευή επιδέχεται σήμανση ΕΚ. Επόμενη διαφάνεια. This shows ε, ευρύτατο λοιπόν φάσμα προϊόντων, το βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, από πολύ μεγάλα μέχρι πολύ μικρά, ε, ε, επί παραγγελία, αλλά όχι, χαλίβδινες γέφυρες, κτίρια, αποθήκες. Αν καταρρεύσει οτιδήποτε από αυτά θα είναι καταστροφικό από πλευράς απώλειας σεζόν και από πλευράς οικονομικών ζημιών. Θα μπορούσατε να πάτε πίσω στην προηγούμενη διαφάνεια σας παρακαλώ. Ε, πάνω πάνω εκεί που λέει δομικά υλικά. Ε. Uh, right. There's a hyperlink there, I think. Well, there was a hyperlink. Okay, never mind. Well, I was going to show you and it's... Ε, ήθελα να σας δείξω κάτι. έχετε στους φακέλους σας ε, την πρώτη χαλίδινη γέφυρα που έλαβε σήμανση στην Ιρλανδία. Ε, είναι μία ε, κρεμαστή γέφυρα του 1911. Την κατεβάσαμε, την ε, ανασκευάσαμε, την ανεγύραμε και ε, υπάγεται τώρα στην οδηγία περισήμανσης ΕΚ και τι γίνεται τώρα που θα υπάρχουν οι δύο οδηγίε, θα επιδέχονται σήμανση ΕΚ δυνάμει και των δύο διαφορετικών οδηγιών. τι πιστεύουμε εμεί για τη σήμανση ΕΚ. Ε, υποστηρίζουμε τον ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα της ε, σήμανσης για προϊόντα κέρυας σημασίας. Θα θέλαμε αυτό να ισχύει σε ολόκληρη την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα που κατασκευάζουμε. Θεωρούμε ότι με τη σήμανση θα αναβαθμιστεί η ποιότητα και ο επαγγελματισμός του κλάδου τα χαλίδινα προϊόντα όπως η δοκή ε, και άλλα, για άλλες δομικές κατασκευές, ε, πλαίσια, οι κρυώματα, ε, θα υποφεληθούν από τη νέα σήμανση. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις εδώ και χρόνια, ώστε να έχουμε τα απαιτούμενα συστήματα, ανθρώπους και κατάρτιση για να επιθέτουμε την σήμανση βάσει των ακανονισμών που αναμένεται να εγκριθούν σύντομα Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που κατασκευάζουμε εμεί και άλλα κατασκευαστικά προϊόντα. Είναι safety critical. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι κρίσιμο, να, είναι κέρια σημασία να είναι ασφαλή. Όπως ε, τα γέφυρε, παραδείγματο χάρη, είναι μεγάλα προϊόντα, είναι τεράστια προϊόντα ε, και έχουν πολύ μεγάλο κύκλο ζωής. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δημιουργούν δυσκολίες ε, με τη σήμανση. Ευτυχώς είναι υποέλεγχο. Αυτά ε, τα προϊόντα δεν πρέπει να υπαχθούν στην εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 5 κατά τη γνώμη μας. Ε, οι χαλίδινες ε, γέφυρες και οι, οι ουρανοξύστες υποθέτω και εσείς δεν θα θέλετε να υπαχθούν σε αυτή τη δυνατότητα απόκλησης και όπως και οι προλαλήσαντες νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλύτερους ορισμούς. Ένα θέμα ε, είναι πού ε, θα επιθέσει κανείς τη σήμανση. Τρία σημεία προβλέπουν στον κανονισμό πάνω στο προϊόν, αλλά με μεγάλο πού θα το βάλετε. Στη συσκευασία, δεν υπάρχει για τη γέφυρα συσκευασία, ε, για, στην εμπορική τεκμηρίωση, για την υγεία και την ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτό θα πάει στον πελάτη και ίσως εκεί θα ήταν ε, ε, ο καλύτερος ε, τόπος εναπόθεσης της ΣΥΜΑΣ. Επόμενη διαφάνεια, για πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρηθεί η τεχνική τεκμηρίωση. Σε προηγούμενα σχέδια του κανονισμού έγινε η πρόταση να παραμένει η τεκμηρίωση για τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Μα αυτό μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Οι υπεραγορές, 25 χρόνια κύκλο ζωής, 60 χρόνια για τα η οι γέφυρες 125 χρόνια. Σαφέστατα Πολλέ κατασκευαστικές εταιρείε θα έχουν κλείψει μέχρι να ε, κλείψει για το προϊόν οπότε ε, ο κατασκευαστής ε, ευτυχώς τελικά θα υποχρεούται να διατηρεί την τεκμηρίωση 10 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο 12 γιατί είναι νομοθετική, δεν είναι δημόσιο έγγραφο το πολιτήριο συμβόλαιο οπότε πρέπει να διατηρηθεί. Ε, και η σήμανση ΕΚ θα αποκτήσει νέα σημασία. Ε, αρχίζουμε να συλλέγουμε χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν μόνο και μόνο για την αρχική θέση σε εμπορία, όχι για να αποφασίσει ο κατασκευαστής αν, θα, αν πληρεί ε, τις προϋποθέσεις το προϊόν, αλλά εισαγάγουμε και την έννοια της βιωσιμότητας. Και γι' αυτό πρέπει να διατηρούμε την τεκμηρίωση για ολόκληρο τον κύκλο ζωή του προϊόντο. Βιωσιμότητα λοιπόν, για να ε, μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε και να επαναχρησιμοποιήσουμε το προϊόν μετά ε, το πέρασε του ε, κύκλου ζωή του. Και ποιο θα το κάνει αυτό, μάλλον ο ιδιοκτήτη. Για την εξαίρεση τώρα όπως και οι συνάδελφοι θα συμφωνήσω ότι την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτά που κατασκευάζουμε κατασκευάζονται επί τούτο και άρα θα πρέπει να ε, υπαχθούν στην εξαίρεση. Όχι, διαφωνώ. Για λόγους ε, δημόσιας ασφάλειας ε, και επειδή είναι κέρια σημασία να είναι ασφαλή χρειάζεται σύστημα ελέγχου πιστοποίησης ούτως ώστε να μεριμνήσουμε για την ασφάλεια των προϊόντων δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε την ασφαλή για δημόσια χρήση. Σα ε, σας μίλησα για την βιωσιμότητα, είναι η έβδομη βασική απέτηση έργων. Ε, τι είδους πράγματα θα πρέπει να δηλώσουμε στην, ε, στο χαλιβουργικό κλάδιο. θεωρούμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για την ενέργεια, δηλαδή πώς ενέργεια δαπανούμε για να φτιάξουμε ένα κομμάτι χάλιβα. Επίσης το, το κομμάτι που πάει για ανακύκλωση, οποιοδήποτε χαλιβουργικό προϊόν κανονικά ε, οδηγεί εν μέρη σε ανακύκλωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 60% των προϊόντων ανακυκλώνονται. Ε, είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση. Ορισμένες φορές κατεδαφίζουμε τα κτίρια και τα ανεγείρουμε και πάλι. Αναρωτιέμαι πώς θα λειτουργήσει αυτό στον κανονισμό. Ε, το ένα εκατομμύριο λίρες δαπανώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο όχι για τα πλαίσια αλλά για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων ε, και προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση των ε, χαλιβουργικών αυτών ε, πλαισίων το 2050. Ε, για τη σήμανση έχουμε κάνει διάφορες διανοητικές ασκήσεις, ε, δηλαδή πώς να επαναχρησιμοποιήσουμε δομές, κατασκευές ε, που κατασκευάστηκαν το 50 ή το 60, πριν αρχίσουν να ισχύουν οι κανονισμοί, πριν προκύψει καν η σήμανση έκτοτε. Δεν είχαν πολλές πληροφορίες για τις διαστάσεις, για τις ιδιότητες, για τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν την χαλίδινη κατασκευή. Οπότε τι κάνουμε για να βρούμε τους φακέλους και να έχουμε τα στοιχεία για να κάνουμε τη σήμανση. Τέτοιου πράγματα πρέπει να μας ε, προβληματίζουν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιθέσουμε τέτοια σήμανση ε, ε, σε αυτά τα προϊόντα, τα προϊόντα που κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται στα νέα κτίρια. Αυτά αντίθετα επιδέχονται σήμανση βάσει του νέου κανονισμού. Είναι η Πρώτη τελευταία μου διαφάνεια για την αστυνόμευση. Ο κλάδο ανησυχεί γι' αυτό. Ε, ε, ανησυχούμε ότι θα υπάρξουν ε, κατασκευαστικέ εταιρείε που δεν θα συμμορφωθούν ε, με τις νομοθετικές διατάξεις και θα ε, επιθέσουν πλαστή σήμανση. Και ανησυχούμε ότι οι αρχές δεν έχουν επαρκείς πόρους για να αστυνομεύουν την κατάσταση, να επιβλέπουν την κατάσταση. Ε, τα πρότυπα εμπορικών συναλλαγών δεν προβλέπουν να πηγαίνει κανείς από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και να βλέπει αν πληρούνται οι προδιαγραφές της σήμανσης και ο κλάδος μας ε, θα ήθελε να συστήσει ένα ανώνυμο σύστημα προειδοποίησης για να καταγγέλουμε τους, ε, τις κατασκευαστικές εταιρείες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Αλλά χρειάζεται κεντρικό μητρό ε, των κατασκευαστών που χρησιμοποιούν σήμανση έκεντη αυτή περιπτώση. Επόμενη διαφάνεια. συνοπτικά η βιομηχανία μας υποστηρίζει την υποχρεωτική σήμανση ΕΚ e για προϊόντα κατασκευαστικά που έχουν κέρια ε, σημασία ως προς την ασφάλειά τους. Ε, και ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί για 10 χρόνια ή και περισσότερο η τεχνική τεκμηρίωση, κυρίως ως προς τα χαρακτηριστικά για τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Για την επόπτευση, για την αστυνόμευση πρέπει να μας προβληματίσει το θέμα, δηλαδή πώς ακριβώς θα ελέγχουμε τη συμμόρφωση με τη σήμανση ΕΚ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδού, ολοκλήρωσα την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very Σας ευχαριστούμε θέρμα, κύριε Μόρ. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια οδηγία για την Γενική Οδηγία Ασφάλειας Προϊόντων. Και εκεί αναφέραμε το θέμα της αστυνόμευσης. Είναι σημαντικό για να εξασφαλίσουμε εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων. Ο κύριος Κόμανς. Σας ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τη ΦΙΕΚ, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικού Κλάδου, που είναι μια οργάνωση που υπάρχει εδώ και 100 περίπου χρόνια και εκπροσωπεί κατασκευαστές και εργολάβους ε, καθώς και πολιτικούς μηχανικούς 29 χώρες και 34 διαφορετικές ομοσπονδίες κατασκευαστικού κλάδου. Όταν ε, μιλούμε για εργολάβους, καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα εργολάβων. Μιλούμε για τεράστιο αριθμό μικρών ουσιαστικά επιχειρήσεων. Και εγώ είμαι, έχω μια μικρή επιχείρηση, λιγότερο από 100 ανθρώπους, 12 εκατομμύρια τζίρο ετήσιο και εμπίπτωση κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων. 7,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι μικρότερη από τη δική μου και δεν θεωρώ τη δική μου επιχείρηση ιδιαίτερα μεγάλη, ούτε καν μεσαία. Δηλαδή έχουμε 7 εκατομμύρια, 5 ε, εκατομμύρια συγγνώμη αυτοαπασχολούμενους, 2,5 εκατομμύρια πολύ μικρές λιπούτιες επιχειρήσεις που απασχολούν 2 ή 3 εργαζόμενους. Ως εκ τούτου έχουμε 10 με 12 εκατομμύρια ανθρώπους που κάνουν την παραλαβή τέτοιων δομικών προϊόντων στα εργοτάξια. Και εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για τους καταναλωτές τέτοιων προϊόντων δόμησης, γιατί το επίπεδο μόρφωσης αυτών των ανθρώπων είναι αντίστοιχο του επίπεδου μόρφωσης ε, των ανθρώπων που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν ένα λίγο τυρί ή μια σοκολάτα. Είναι σημαντικό αυτό όσο όταν συζητούμε για δύο πολύ κέρια ζητήματα. Το πρώτο είναι η διευκρίνηση του πεδίου εφαρμογή της ρύθμιση. Μιλούμε δηλαδή για προϊόντα και κατασκευαστές και όχι για εργολάβους. Και για τους ε, εργολάβους είναι σημαντικό να έχουμε ε, λεπτομεριακές και αξιόπιστες πληροφορίες για το προϊόν. Τι σημαίνει αυτό. Όταν κανείς παραλαμβάνει ένα προϊόν σε ένα εργοστάσιο θα πρέπει ε, να μπορεί με μια ματιά να καταλαβαίνει γιατί προϊόν πρόκειται και να βλέπει και το σήμα ΕΚ. Δεν χρειάζεται να πρέπει να διαβάσει μια εκτενέστατη δήλωση για να δει τι προϊόν παραλαμβάνει. Επίσης, ο εργολάβος που είναι ο καταναλωτής αυτού του προϊόντο, θα πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει ότι φτάνει στο εργοτάξιο το προϊόν και μάλιστα να μπορεί να εντοπίζει το προϊόν χωρίς καμία αμφισημία. Να μην χρειάζεται να ψάξει έναν ιστότοπο ή σε μια ιστοσελίδα για να καταλάβει ποιο, για ποιο προϊόν πρόκειται. Και όταν τα προϊόντα φτάνουν στο εργοτάξιο θα πρέπει να έχουν επαρκή πληροφόρηση αλλά όχι ε, υπερβολική ώστε να δημιουργείται σύγχυση για το προϊόν. Σε ό,τι αφορά το σήμα καταλάβετε ότι πρόκειται για κάποιες ε, ε, ενδείξεις που αναφέρει ότι είναι για, για εσωτερική χρήση. Ε, για, για παράδειγμα, για κεραμίδια. Αν λέγεται κεραμίδια προορίζεται για εσωτερική χρήση, φυσικά κάποιος που θέλει να βάλει κεραμίδια ή τούβλα στην πρόσωψη θα πρέπει να τηλεφωνήσει για να ρωτήσει τι εννοείται εσωτερική χρήση, δεν μπορούμε δηλαδή να τα βάλουμε στην, στην πρόσωψη. Επίσης, αν στο προϊόν βλέπουμε μόνο μία ηλεκτρονική διεύθυνση ή ένα κωδικό, είναι δύσκολο να καταλάβουμε για τι προϊόν πρόκειται. Γι' αυτό συμφωνούμε με την πρόταση του Συμβουλίου και το άρθρο 9 που μιλάει για επαρκείς πληροφορίες σε περίπτωση που γίνεται παραλαβή προϊόντων δόμησης στο εργοτάξιο. Θα πρέπει το σήμα ΕΚ να δίνει αρκετές, επαρκείς μάλλον πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν. Σε ό,τι αφορά την διευκρίνηση του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού, θα ήθελα να πω ότι και πάλι μιλούμε κυρίω για το άρθρο 5. Το έγγραφο μιλά για κατασκευαστές και για προϊόντα που τίθενται στην αγορά, που διατίθενται στην αγορά. Όταν αρχίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο 5, διαπιστώνουμε ότι προβλέπει και εξαιρέσεις. Το σημείο α, το εδάφιο α του άρθρου 5 μιλά για εξαιρέσει ε, κατασκευαστών που εγκαθιστούν προϊόντα. Ένας κατασκευαστής όμως που εγκαθιστά προϊόντα σε εργοτάξιο είναι πια εργολάβος, δεν είναι κατασκευαστής. Όταν ε, ο εργολάβος ουσιαστικά προκατασκευάζει ένα δόκο, μια δόκο στο, είτε στο εργοτάξιο είτε στην αποθήκη του, ουσιαστικά εκτελεί το, το έργο για το οποίο έχει προσληφθεί. Όταν όμως ο ίδιος εργολάβος, αντί να χρησιμοποιεί αυτό το δοκό που κατασκεύασε, το πουλάει, κατασκευάζει 100 και πουλάει σε άλλους, τότε γίνεται κατασκευαστής. Θα πρέπει η διάκριση να είναι σαφής. Κάποιος που εσωματώνει ένα προϊόν σε ένα κτίριο είναι εργολάβος. Κάποιος που κατασκευάζει αυτό το προϊόν και το παραδίδει σε ένα εργοτάξιο είναι κατασκευαστής. Ως εκ τούτου, οι η εξαίρεση του σημείου α δεν ισχύει πια, γιατί η εξαίρεση αυτή μιλά για δραστηριότητες αργολαβίας, ε, για δραστηριότητες του εργολάβου, Σε ό,τι αφορά το εδάφιο β του άρθρου 5, φαίνεται ότι καλύπτει την περίπτωση όπου σε ένα εργοτάξιο τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά, ορισμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Και πάλι όμως αυτή η δραστηριότητα είναι δραστηριότητα κατασκευαστή και όχι εργολάβου. Αν για παράδειγμα αγοράζω ένα λούκι που είναι κατασκευασμένο από ε, αυτό το λούκι ως προϊόν ε, θα πρέπει να φέρει το σήμα ΕΚ. Όταν όμως εγώ τροποποιώ αυτό το ε, λούκι στην εσωμάτωσή του στην αγορά, στο εργοτάξιο που δουλεύω, τότε το σήμα ΕΚ δεν ισχύει πια, γιατί εγώ το έχω τροποποιήσει. Αν επίσης ε, αγοράσω κάποια λούκια και δεν μπορώ να τα ταιριάξω και απλώς τροποποιώ ελαφρώς, τότε δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις, Κατά τη γνώμη μου λοιπόν το σημείο Β του 5 δεν έχουν νόημα γιατί αφορά, αφορούν περισσότερο εργολαβικές δραστηριότητες και όχι κατασκευαστικές. Επίσης αν κατασκευάσει κανείς μια γέφυρα δεν θα χρειάζεται να βάλει και το σήμα ΕΚ. Τώρα, αν κανείς κατασκευάζει τη γέφυρα σε, μια αποθήκη, σε ένα εργαστήριο 100 χιλιόμετρα από το σημείο που θα την τοποθετήσει ή στο σημείο που θα την τοποθετήσει δεν έχει δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει διαφορά. Αυτός που κατασκευάζει τη γέφυρα είναι κατασκευαστής. Γιατί θα κατασκευάσει 25 γέφυρες και θα τις πουλήσει σε 25 διαφορετικούς εργολάβους που θα τις εγκαταστήσουν. Όπου και να κατασκευάζονται οι γέφυρες είναι άσχετο με το χαρακτηρισμό του κατασκευαστή. Επίσης ζητήσαμε σαφήνεια στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Οι εργολάβοι δεν είναι κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές ε, είναι αυτοί που εμπίπτουν στην, ε, στον κανονισμό. Οι εργολάβοι αγοράζουν προϊόντα που έχουν το σήμα ΕΚ. Δεν κατασκευάζουν προϊόντα που θα πρέπει να φέρουν το σήμα ΕΚ. Επίσης, ο κανονισμός θα πρέπει να περιορίζει τον αριθμό των ε, πληροφοριών που, που προβλέπονται σε άλλες νομοθετικές διατάξεις για τα προϊόντα. Αν θέλετε άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτά που σας είπα, μπορείτε να κοιτάξετε το site μας fiec.eu. Σας... ευχαριστούμε. Ο καθηγητής Μπόσενμαϊερ τώρα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα αλλάξω σε μεγάλο βαθμό αυτά που είχα σκοπό να πω, διότι επαναλάβω πολλά από αυτά που ήδη υπόθηκαν. Πρόκειται για επικρίσεις τις οποίες είχα σκοπό να επαναλάβω, τις ακούσαμε όμως ήδη. Και άλλωστε σας έχω υποβάλει και μία γνωμοδότηση στα αγγλικά. Παρακαλώ να τη διαβάσετε. Εκεί περιέχονται όλα αυτά. Κυρία Πρόεδρε, είπατε κάτι νωρίτερα, το οποίο Ευχαριστώ ακούμε όσον αφορά τα Eurocodes. Μας είπατε ότι θα βρίσκεται συναρπαστικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου λέγοντας ότι ένα από τα βασικά προβλήματα το και αυτό είναι γνωστό, είναι ότι οι κανόνες υπολογισμού για, τα, για τις κατασκευές δεν μπορούν να εναρμονιστούν και δεν έχει νόημα να... είναι πρόβλημα η εναρμόνιση των προϊόντων εφόσον δεν είναι εναρμονισμένοι και οι άλλοι κανόνες. Κατά την εφαρμογή και αυτού του κανονισμού θα υπάρχουν τα ίδια προβλήματα διότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον τρόπο υπολογισμού, τους κανόνες υπολογισμού. Και έχουμε 350 κανόνες ε, οι οποίοι είναι λίγο πολύ έτοιμοι ε, που έχουν να κάνουν με την ε, αηφορία. Και γιατί, όχι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να είναι όλα εναρμονισμένα, αλλά δεν γίνεται στην πράξη να μην υπάρχει αυτή η εναρμόνιση. Δεν θα είναι πλήρης η, δήλωση του επισήμανση του προϊόντος εάν δεν ληφθούν υπόψη χίλιοι ε, ε, ε, παράμετροι που είναι Χίλιες παράμετροι που ε, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Από ό,τι κατάλαβα, μας ζητάτε να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας. Ε, γι' αυτό θα εκφράσω και εγώ τη δική μου επιθυμία. Θα παρακαλούσα τα κράτη-μέλη μέσω πρόθεσμα να εναρμονίσουν τους κανόνες αυτούς για να πετύχει καλύτερη η εναρμόνιση που αφορά τα δομικά υλικά. Θα είμαι σύντομος όσον αφορά την ε, αδειοδότηση. Εργάζομαι με το θέμα αυτό πολλά χρόνια. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Κούπερ. Εάν μου επιτρέπετε θα αναφέρω ότι Είναι απαραίτητες ε, αυτές οι ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ε, και στο, στην παγκόσμια αγορά, διότι είναι επιθυμητές στον διεθνή ανταγωνισμό. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι Στην ΕΟΤΑ χρειάζεται μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Το είπε ήδη ο κύριος Κούπερ και συμφωνώ ε, για τα EAD, για τις ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις οι οποίες αποτελούν την βάση για τις άδειες που εκδίδονται θα πρέπει να έχουμε εμπειρογνώμονες από τις, τους διάφορες φορείς έγκρισης και η χρηματοδότηση θα πρέπει να σέβεται τον, ε, την αρχή της ουδετερότητας, θα πρέπει δηλαδή σε μεγάλο βαθμό να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίζεται η αυτονομία του φορέα. Τα ETA οι ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις χρηματοδοτούνται από μόνες τους. Ε, αυτή τουλάχιστον ε, είναι η εμπειρία μας στη Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτό, να επαναλάβω την έκκλησή μου. Στη θέση του Συμβουλίου έχει διορθωθεί κάπως η κατάσταση. Στο παρελθόν πάντα είχα το άγχος ότι οι άδειε, οι εγκρίσει δεν μπορούν να αποτελέσουν δεύτερη ε, οδό. δεν θα ήθελα το CEN να ε, χειρίζεται και τα καινοτόμα προϊόντα, διότι η επισήμανση μπορεί να γίνει μόνο για προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά, τα οποία είναι χρήσιμα και έχουν αποδείξει την αξία τους. Χρειαζόμαστε την ε, διαδικασία αδειοδότησης για τα καινοτόμα προϊόντα ε, ως πρόλογο στην εισαγωγή για ε, πριν τη διάθεση στην αγορά. Τα specific technical documentations είναι πολύπλοκα έγγραφα αναφέρονται στους ε, απλοποιημένους αυτούς κανόνες, δεν ορίζονται όμως. Ε, αναφέρεται λίγο χαλαρά ότι εντάξει, ας εκπονείτε τότε ένα STD. Δεν ξέρω αν φταίει που είμαι κάπως ηλικιωμένο. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, μου φαίνεται αστείο να λέει κανείς «Ε, ε εντάξει, φτιάξε ένα STD χωρίς να ορίζεται τι ακριβώς είναι αυτό». Τα προϊόντα αυτά ε, συμμετέχουν στον ανταγωνισμό, θα πρέπει να είναι και ασφαλή. Επιτρέψτε μου να ε, κάνω την εξή παρατήρηση. Ο τομέας μου είναι τα έγγραφα που έχουν να κάνουν με την δήλωση απόδοσης. Στο άρθρο 6 αναφερόμαστε στην πληρότητα της επισήμανσης, της δήλωσης του προϊόντος. Από ό,τι κατάλαβα από τους προλαλήσαντες, αν έχω 10 χαρακτηριστικά και για ένα χαρακτηριστικό, επειδή μου φαίνεται πολύ βολικό και πιο φθηνό ε, να πω ότι δεν ε, χρειάζεται εδώ ε, δήλωση απόδοσης. Ε, αυτό οδηγεί σε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, για το πάχος ε, ενός τούβλου, επειδή είναι εύκολο να το μετρήσω, ε, αναφέρω το χαρακτηριστικό, για τα άλλα επειδή είναι πιο δύσκολο να υπολογιστούν, δεν γράφω τίποτα. Μας ενδιαφέρει η ομοιογένεια μιας αγοράς Ε, πώς ε, θα κρίνω εγώ, πώς θα αξιολογήσω εγώ ένα προϊόν το οποίο παραδίδεται στο εργοτάξιο. Το βλέπω μεν, αλλά δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι γίνεται με το προϊόν αυτό. Πρέπει να το στείλω πίσω. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να υπάρχει εδώ κανόνας. Από ό,τι κατάλαβα από την Κομισιόν και εκείνη θεωρεί ε, απαράδεκτη την κατάσταση και πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Δεύτερη παρατήρηση, προσαρμογή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα προϊόντα. Θα πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς, και δεν είναι πάλι γερμανική ιδιαιτερότητα αυτό, πρέπει όλοι να το κάνουν αυτό, διότι δεν υπάρχουν ακόμα ενιαίοι κανόνες υπολογισμού στον τομέα αυτών. Καταλήγω λοιπόν σε μια συγκεκριμένη αξία ε, εξετάζοντας μια συγκεκριμένη προδιαγραφή και εφαρμόζω τις γερμανικές προδιαγραφές θα πρέπει να έχω έναν πίνακα αντιστοιχίας ε, που να δείχνει τον, ε, την δήλωση απόδοσης ε, με τους εθνικούς κανόνες. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουμε έτσι. Θα πρέπει όμως να κάνουμε κάτι διότι το ίδιο θα ισχύει και στα άλλα κράτη-μέλη. Εποπτεία της αγοράς, ναι, ε, λείπει εδώ. Ένα προϊόν που δεν έχει δηλωθεί είναι αδύνατον να ελεγχθεί στην αγορά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν ο φορέας εποπτείας της αγοράς ε, ζητήσει επανεξέταση των ε, δηλώσεων απόδοσης που λείπουν. Αλλά έτσι αυξάνω τη γραφειοκρατία, ε, επιβάλλω δαπάνες στον κατασκευαστή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το άρθρο 6 λοιπόν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Τα, οι άλλες μου δύο παρατηρήσεις είναι πιο σύντομες. Ε, άρθρο 6, 3, ε. Εδώ κατά τη γνώμη μου λείπει να υπάρχει τρόπος υπολογισμού συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Μιλάμε εδώ για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Θα πρέπει να μπορώ να μετρήσω, για παράδειγμα, την αντοχή ενός προϊόντος. Θα πρέπει να μπορώ να τον υπολογίσω μόνη μου, να μην πρέπει να ε, κάνω επιστημονικές δοκιμές. Αυτά όσον αφορά για παράδειγμα την αντοχή ενός προϊόντος ε, ή την ε, δυνατότητα θερμομόνωσης. Και τέλος, στο 6.3 σίγμα F υπάρχει το No Performance Determined, το NPD. Ενώ οι προδιαγραφές ε, προβλέπουν την συγκεκριμένη κατηγορία, δεν δηλώνεται η απόδοση του προϊόντος. Κυρίες και κύριοι, αυτό κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ρυθμίζεται. Δεν μπορεί απλά ο κατασκευαστής να πει ότι δεν χρειάζεται να, ε, να πει ότι δεν χρειάζεται να το δηλώσω αυτό. Δεν θα πρέπει να είναι προαιρετικό το να μην το δηλώνει. Και τελευταία παρατήρηση, οι κανόνες απλοποίησης. Ξέρω ότι Πολιτικά είναι πολύ ε, ευαίσθητο θέμα αυτό, πολύ λεπτό. Θα πρότεινα να διαγραφούν τελείως τα άρθρα 137 και 138. Κανείς ε, δεν έχει παραπονεθεί μέχρι στιγμής, ε, αλλά μετά τη σημερινή συζήτηση θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να παραπέμπουμε αποκλειστικά στο άρθρο 5. Αλλά, όπως άκουσα σήμερα, θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις στο άρθρο 5, διότι δεν είναι σαφείς οι ορισμοί. Αυτό σημαίνει ότι την διαδικασία στα άρθρα 37 και 38 που έχουν γραφεί με πολύ καλές προθέσεις, ε, την απλοποίηση της νομοθεσίας, ε, τη μείωση του κόστους, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Αλλά η διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 37 και 38 δεν ε, είναι καθόλου παρόμοιες με αυτές στα άρθρα 3 με 6. Οι ορισμοί εδώ είναι ατελείς και λάθος θα πρέπει να διορθωθούν. Βλέπουμε σημαντική στρέβλωση της αγοράς και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και κλείνω, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, στο άρθρο 37 αποτελούν το, αντιπροσωπεύουν το 4% των, ε, ε, των προμηθευτών. Πώς θα δικαιολογούσαμε μια τέτοια, μια τέτοια διάλυση του όλου συστήματος ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Μάικλ Ρόμπερτς από την ΚΑΝ. Um, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ονομάζομαι Μάικλ Ρόμπερτς και εκπροσωπώ την Επιτροπή για την ε, ε, ασφάλεια στον χώρο εργασία, την υγεία και την προτυποποίηση από τη Γερμανία. Θα σας παρουσιάσω τη γνώμη της Επιτροπής μας και θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ΚΑΝ, που είναι μια τριμερή οργάνωση στη Γερμανία, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, εκπρόσωποι των εργοδοτών και εκπρόσωποι των κρατικών αρχών. Από τις συζητήσεις που κάνουμε στην ΚΑΝ, την Επιτροπή μας, καταλήγουμε σε μία γνωμοδότηση που είναι η κοινή γνωμοδότηση των τριών μερών που συναποτελούν την ΚΑΝ και είναι ουσιαστικά η επίσημη γνώμη, η επίσημη θέση της Γερμανίας για την πρωτοτυποποίηση. Το θέμα της προστασία των προϊόντων, της ασφάλειας των προϊόντων μάλλον για τα δομικά προϊόντα είναι πολύ σημαντικό θέμα και μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό, γιατί από καιρούς καιρό είχαμε περιπτώσεις προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την εντύπωση που έχουμε για το πώς θα πρέπει να είναι ένα ασφαλές προϊόν. Σε ό,τι αφορά τα δομικά προϊόντα, βλέπετε στη διαφάνεια ότι έχουμε ένα ευρύτατο φάσμα τέτοιων προϊόντων δόμησης. Έχουμε από ένα ε, σακί τσιμέντου, ε, έχουμε σωλήνες, δοκούς, πατώματα, μονοτικό υλικό, μηχανήματα, περιστεφόμενες πόρτες, ε, εξοπλισμό υψηλής πίεσης, μια ευρύτατη γκάμα λοιπόν προϊόντων. Όλα αυτά τα προϊόντα θεωρούνται προϊόντα δόμησης. Και όταν μιλούμε για προϊόντα δόμησης, μιλούμε για έναν τεράστιο κλάδο βιομηχανικής παραγωγής. Και αυτός ο κλάδος, κατά τη γνώμη μα έχει το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή του και να και διεκδικεί μία σωστή, περιεκτική, πάγια και δίκαιη ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ασφάλεια των προϊόντων, κάτι που δεν ε, έχει καλυφθεί από τις μέχρι τώρα οδηγίες ή στα έγγραφα του Συμβουλίου για τον κανονισμό. Κάτι που δεν θα πρέπει να εμπίπτει στη ρύθμιση, κάτι που δεν θα πρέπει να διαθετείτε, Γιατί υπάρχουν κάποιε διατάξει που μιλούν για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον χώρο εργασία. Υπάρχουν όμω άλλα νομοθετικά κείμενα γι' αυτό. Και το λέω γιατί πολύ συχνά οδηγούμαστε σε σύγχυση, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να ρυθμίσει τα πάντα, ό,τι συμβαίνει δηλαδή σε, ενεργοτάξιο. σε Αυτό δεν ισχύει, γιατί ε, το θέμα της ασφάλειας και της υγείας ε, σε ενεργοτάξιο, εργοτάξιο, για παράδειγμα, εμπίπτει στην Εθνική Νομοθεσία και δεν έχει καμία σχέση με τον κανονισμό CPR, τον κανονισμό για τα προϊόντα δόμησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει στον κανονισμό αυτό είναι η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, κάποια στοιχεία της ασφάλειας των προϊόντων και ο κανονισμός αυτός είναι ε, ο μόνος σωστός ε, κανονισμός που θα πρέπει να καλύπτει αυτά τα προϊόντα δόμησης. Επόμενη διαφάνεια. Όταν ε, κοιτάξει κανείς εκ του σύνεγγυ στην παραγωγή των προϊόντων δόμησης διαπιστώνει ότι έχουν ποικίλα χαρακτηριστικά στη διάρκεια της, ε, του κύκλου ζωής τους, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκονται. Έχουμε την φάση της μεταφοράς, ε, τη φάση της, χρημα... της συναρμολόγησης, τη φάση της χρήσης αφού ολοκληρωθεί το έργο στο εργοτάξιο, της εσωμάτωσης ε, σε συγκεκριμένο έργο και έχουμε και τη φάση της συντήρησης όλες αυτές οι φάσεις, όλα αυτά τα διαφορετικά στάδια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλούμε για την ασφάλεια των προϊόντων δόμησης. Η θέση του Συμβουλίου για τον κανονισμό αυτό δυστυχώς μιλά μόνο για την υγιεινή και την, την υγιεινή και την υγεία των κατοίκων και των γειτόνων. Όχι όμως για την υγεία των εργαζομένων. Δεν εξετάζεται παρκώς το θέμα αυτό στη θέση του Συμβουλίου. Αν ρίξουμε μια ματιά σε στατιστικά στοιχεία, θα δούμε ότι η πλειοψηφία των ατυχημάτων που αφορούν κατά κάποιο τρόπο την ασφάλεια των προϊόντων δεν γίνονται κατά τη φάση της χρήσης των προϊόντων σε προηγούμενες φάσεις που ανέφερα προηγουμένως. Οπότε αν δεν θεσπίσουμε διατάξεις για τις φάσεις αυτές, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο νομοθετικό κενό στον οικονομισμό. Είναι αναφυσβήτητο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ένα ασφαλές προϊόν είναι το σημείο κλειδί για να μειωθεί το ποσοστό ατυχημάτων στα εργοτάξια. Ε, δυστυχώς ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους κλάδους με το υψηλότερο ποσοστό ή ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων στο χώρο εργασίας. Και από γερμανικές στατιστικές ε, ε, πληροφορίες ξέρουμε ότι ο αριθμός των ατυχημάτων στο κατασκευαστικό κλάδο είναι τριπλάσιος από τα ατυχήματα σε άλλους τομείς. Και αυτό πολλές φορές οφείλεται σε προϊόντα που δεν είναι ασφαλή. Ένα τμήμα όμω, ε, βέβαια των ατυχημάτων οφείλεται στην ασφάλεια των προϊόντων. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα προϊόντα για τα ατυχήματα αυτά. Πάντω ε, έστω και ένα ατύχημα να αποτρέψουμε εξαιτία της βελτίωση, χάρη στη βελτίωση των προϊόντων και αυτό αξίζει. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα τη ασφάλεια των προϊόντων δόμηση στον κανονισμό CPR. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε κάποια παραδείγματα. Η ασφάλεια των προϊόντων δόμησης θα πρέπει να εξεταστεί πριν τη φάση της χρήσης τους. Σας μίλησα για ένα προκατασκευασμένο τμήμα που μεταφέρεται, για παράδειγμα. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να το γνωρίζει και να φροντίσει πώς θα μπορέσει αυτό το προϊόν που μεταφέρει να ενσωματωθεί σωστά στο κατασκευαστικό έργο. Επίσης, μπορούμε να έχουμε μια ασθένεια εξαιτία υψηλή περιεκτικότητα χρώμιου στο τσιμέντο. Πολλέ φορέ είχαμε τέτοιε περιπτώσει Εμφάνιση κρουσμάτων ή ακόμη και εγκαυμάτων εξαιτία τη υψηλότερη περιεκτικότητας ε, χρωμίου ή, άλλου, ουσία σε ένα σωματωμένο προϊόν. Τέτοιου είδους ε, θέματα ασφάλειας θα πρέπει να διαθετηθούν και να ρυθμιστούν σε επίπεδο προϊόντος. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε μία περίπτωση ασφάλειας στη διάρκεια της ε, φάσης χρήσης ή της φάσης συντήρησης για παράδειγμα κάποια στοιχεία της ε, ε, διόρθωσης της ε, σκεπής έπεσε στο πάτωμα και γλίστρησε ο εργαζόμενος ε, και είχαμε μια τέτοια περίπτωση εργασιακού ατυχήματος. Αν το προϊόν ήταν ασφαλέστερο δεν θα γινόταν, ε, θα αποφεύγουμε το ατύχημα ή αν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες πάνω στο προϊόν θα είχε αποφευθεί αυτό το ατύχημα. Αν λοιπόν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κατασκευαστή να παράγει ασφαλέστερα προϊόντα, αυτό θα βοηθούσε και την καλύτερη χρήση και σωμάτωσή τους. Ένα άλλο πρόβλημα που οφείλεται στον αμίαντο. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της ε, χρήσης ε, ενός προϊόντος, χρειάζεται μερικές φορές να, να καταδαφίσουμε το κτίριο εξαιτία ε, προβλήματος υγείας, όπως συνέβη με τον αμίαντο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Κατά τη γνώμη μας υπάρχει ένα νομικό κενό στον κανονισμό προϊόντων δόμησης. Θα πρέπει αυτό το κενό να γεφυρωθεί. Αναφέρθηκε το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει μεγάλο βαθμό προστασίας για την ασφάλεια και την υγεία. Δυστυχώς ε, αυτή η απέτηση του άρθρου 114 δεν ε, πληρείται στον κανονισμό CPR για τα προϊόντα δόμηση. Αυτό το νομικό κενό που δημιουργήθηκε στον κανονισμό θα πρέπει να πληρωθεί. Θα πρέπει να προβλέψουμε και κάποιες ε, διατάξεις ασφάλειας των προϊόντων στις βασικές διατάξεις. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα επιβαρύνουμε με περισσότερη γραφειοκρατία τους κατασκευαστές. Αντίθετα, ουσιαστικά θα είναι ένα εισιτήριο εισόδου της ε, διαδικασίας προτυποποίησης. Και όσοι γνωρίζουν τη διαδικασία προτυποποίησης και ξέρουν πώς λειτουργεί, ξέρουν ότι υπάρχει μια, επιτροπή προτυποποίησης που απαρτίζεται από συγκεκριμένο αριθμό μελών που εκπροσωπούν τους ενδιαφερόμενους. Συνήθως είναι κατασκευαστές. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι κάθονται και συζητούν τις διάφορες πτυχές του προϊόντος και κατόπιν, αφού παρουσιάζεται το θέμα από διάφορες πλευρές, η Επιτροπή συζητά και καταλήγει σε μία απόφαση αν είναι πιστικά τα επιχειρήματα για ένα προϊόν, τα δέχονται, και δίνουν το πιστοποιητικό προτυποποίησης. Αν το επιχείρημα δεν τους πείθει, δεν θα το δεχτούν. Χρειάζεται συνένεση στην Επιτροπή Προτυποποίησης για να περάσει το προϊόν στο επόμενο στάδιο και να λάβει την έγκριση των τεχνικών προτύπων. Οπότε είναι σημαντικό αυτό και για τους κατασκευαστές. Τέλος, μια σαφής διαδικασία θα συμβάλλει και σε αποκατάσταση του ισότιμου και θεμητού ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιου είδους σαφείς προδιαγραφές ασφάλειας είναι εποφελής για όλους, γιατί ο κατασκευαστής και χρόνο και χρήμα για να παραγάγει ένα ασφαλές προϊόν. Πολλές φορές όμως, ε, ε, ακριβώς επειδή μπήκε στον κόπο και έκανε, αφιέρωσε μεγάλο χρόνο και χρήμα, πολλές φορές δεν προλαβαίνει και είναι λιγότερο ανταγωνιστικός από τους ε, υπόλοιπους ανταγωνιστές. Κάτι που είναι απαράδεκτο γιατί ουσιαστικά τιμωρούμε τον πιο έντιμο κατασκευαστή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε για όλους σαφείς προδιαγραφές ασφάλειας προϊόντων προκειμένου να προστατεύσουμε και την ευρωπαϊκή αγορά από έξω κοινοτικού παραγωγούς που ίσως είναι πιο αδίστακτοι. Πού βρισκόμαστε τώρα λοιπόν. Η ασφάλεια των προϊόντων για όλες τις φάσεις ε, του κύκλου ζωής των προϊόντων είναι κάτι που περιλαμβάνεται στη θέση του κυκλου των Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε στην πρώτη ανάγνωση 24 Απριλίου του 2009 και περιλαμβάνεται στο σχέδιο σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση τη θέση του Συμβουλίου. Δυστυχώ όμω δεν περιλαμβάνεται στη θέση του Συμβουλίου όπως έχει διαμορφωθεί. Γι' αυτό ζητούμε επίμονα από την Επιτροπή σας να εμείνει στη θέση που έχει οθετήσει μέχρι στιγμής για το θέμα αυτό και να συμπεριλάβει και προδιαγραφές ασφάλειας προϊόντος στον κανονισμό για τα προϊόντα δόμησης. Μόνο έτσι θα φτάσει αυτός ο κανονισμός στο σωστό επίπεδο εφάμιλο με άλλων οδηγιών και κανονισμών γιατί όπως σας είπα αυτή τη στιγμή η θέση του Συμβουλίου υστερεί σε σχέση με την πρόταση του Κοινοβουλίου και δημιουργεί ένα μεγάλο νομικό κενό. Πιστεύουμε ότι αυτό το κενό θα πρέπει να συμπληρωθεί χάρη της ασφάλειας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα που και που εδώ και χρόνια περιμένουν ένα τέτοιο βήμα και μια τέτοια χειρονομία και μια βελτίωση του κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές ε, για τις ε, κατατοπιστικότατες παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε την ε, Προεδρία, τον εκπρόσωπο της Βελγικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε κάποια σχόλια και εσείς αν θέλετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους εκτός από την τελευταία παρουσίαση Νομίζω ότι η πλειοψηφία υποστηρίζει τις αδρές γραμμές του σχεδίου του Συμβουλίου ε, και κάποιες επιθυμίες ως προς προσαρμογές που μπορούν να γίνουν. Θα ήθελα, εφόσον μου δώσετε το λόγο, να σχολιάσω κάποια ζητήματα. τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας ε, έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία, όπως σωστά είπατε. Όμως, αντίθετα από αυτά που είπατε, το Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτές τις πτυχές και γνωρίζει ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση μέσω της αρχής επικουρικότητας να κατοχυρώσουν όλο αυτό το κομμάτι που σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια. Αυτό το έγγραφο σχετίζεται με τη θέση σε εμπορία των προϊόντων. Δεν είναι σε τέτοιου είδους ε, νομική πράξη που πρέπει να καλύψουμε όλο αυτό το ευρύτατο φάσμα ε, τεχνικών πτυχών και δεν τις εξαντλήσαμε κιόλα σήμερα. Ε, θυμηθείτε ότι υπάρχει μια ε, ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε ένα προϊόν και στη χρήση του και όπως υπενθύμησαν και, άλλες και άλλοι ομιλητές συγγνώμη, το σημαντικό με ένα προϊόν ε, είναι η χρήση του που προβλέπεται από τα κράτη-μέλη με τη δική τους νομοθεσία μέσω της αρχής επικουρικότητας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, ε, ήθελα μόνο ε, να σας πω ότι έχουμε λάβει δεόντως υπόψη αυτή την πτυχή και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τα μέτρα που χρειάζονται. Τώρα, ασχολιάζω και το θέμα των ε, εξαιρέσεων, γιατί αναφέρθηκε από πολλούς ε, ομιλητές και θα ήθελα να προασπιστώ εδώ τη θέση του Συμβουλίου έχουμε προβλέψει εξαίρεση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα ε, μεταξύ άλλων ή μάλλον θα σας πω ότι δεν πρέπει να διαβάζετε μόνο το άρθρο 5 με τις εξαιρέσεις και εδώ απευθύνομαι στον εκπρόσωπο της ΦΙΕΚ ε, για να τον παραπέμψω στους ορισμούς. Ορισμός του παραγωγού, παραδείγματος χάρη, στο άρθρο 2 τον ορισμό της θέσης σε εμπορία και η νομική μας υπηρεσία μας ε, επισήμανε ότι όταν ένας ε, ανάδοχος εργολάβος, κατασκευαστής, ο οποίος όπως θέλετε να τον ονομάσετε, ε, φτιάχνει μία δοκό σε ένα εργοτάξιο ή οτιδήποτε άλλο, η νομική υπηρεσία θεωρεί ότι υπάρχει μεταβίβαση ιδιοκτησίας και άρα θέσει εμπορία. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ε, ο ανάδοχος επομίζεται κάποιες από τις ευθύνες ε, του κατασκευαστή. Γι' αυτό ε, σας μίλησα για το άρθρο 7 ε, τα συστήματα 1, 1 συν και 2 συν, ναι, ναι, εκεί έχουμε προβλέψει εξαιρέσει, αλλά αυτό είναι άλλο διαφορετικό θέμα. Ε, όταν μιλάμε για τις εξαιρέσει ε, του 5α και του 5β, βάση των διευκρινήσεων που ακούσαμε για τη θέση σε εμπορία είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ε, παρεκκλήσεις γιατί αλλιώς θα ανακύψουν νομικά προβλήματα κατά την μεταφορά της ε, νομής ε, του προϊόντος προς τον ανάδοχο και άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε στη θέση σε εμπορία. Αντίθετα, τα προϊόντα, εφόσον χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο εργοτάξιο, δεν θα μεταφερθούν στη συνέχεια και άρα ε, κρίνουμε πως δεν είναι απαραίτητο να φέρουν τη σήμανση ΕΚ και το αναφέρατε κι εσείς. Όταν κατασκευάζουμε κάτι ε, για μια ειδική χρήση, όπως ε, μια γλάστρα, παραδείγματος χάρη, εκεί θα παραμείνει και ε, δεν χρειάζεται να φέρει τη σήμανση γιατί δεν πρόκειται μετά να απολυθεί τα ράφια κάποιου πολυκαταστήματος. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που εκρεμεί, το συζητούμε ακόμη ή ας πω ότι ε, διαφέρει η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη δική μας, είναι το θέμα των μικροεπιχειρήσεων. Τι γίνεται με αυτό το άρθρο 37 που σχολιάστηκε εδώ. Το σχέδιο του Συμβουλίου εν γέννη υιοθετεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τις μικροεπιχειρήσεις και τι προβλέπει αυτή η προσέγγιση λύσεις αρκετά τόσο ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των ε, επιχειρήσεων. Πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, όχι για το 37, αλλά για το άρθρο 36. Να μην χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο STD που ε, χρησιμοποιείται συγκεκριμένα στο άρθρο 37. Μιλήσατε για το άρθρο 37 στην έκθεση που πρέπει να καταθέσει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Ε, νομίζω και ελπίζω πάντως ότι θα μπορέσουν τα μέλη της Επιτροπής σας ε, να συμφωνήσουν με την άποψη του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω και άλλους συναδέλφους. Ε, μήπως Οποιοςδήποτε θα ήθελε να προσθέσει κάτι, ο κύριος Μάιερ. Υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων, αλλά θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση για το άρθρο 6 στους εμπειρογνώμονες, σημείο 3ε. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, γράφει εδώ Γίνεται εδώ αναφορά σε προδιαγραφές ε, στον τόπο στον οποίο θέλει να διαθέσει στην αγορά ο κατασκευαστής το προϊόν. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ο κατασκευαστής παράγει στην, στις Βρυξέλλες, πουλάει σε έναν χονδρέμπορο, ο χονδρέμπορος πουλάει σε λιανοπολιτή. την απόδοση ενός δομικού υλικού, πώς μπορεί να την δηλώσει κάποιος στον τόπο όπου διατίθεται στην αγορά το προϊόν. Για παράδειγμα, εάν το προϊόν στην Ελλάδα ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία ε, ενσωματωθεί σε, κάποιο κτίριο, ε, θα πρέπει να, να ε, ακολουθεί διαφορετικέ προδιαγραφέ, Κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται. Είμαστε σε εσωτερική αγορά. Εφόσον ένα, ε, θα πρέπει ένα προϊόν να έχει άδεια για να πωλείται στην εσωτερική αγορά, και θα πρέπει να υιοθετήσουμε εδώ διατάξεις που να ανοίγουν την εσωτερική αγορά για τα προϊόντα και όχι να ε, υποχρεώνουμε τους κατασκευαστές να πληρούν προδιαγραφές ανάλογα με το πού ε, θα διαθέσουν το προϊόν τους στην αγορά, στη Γερμανία, στην Ελλάδα ή στη Γαλλία. Πιστεύω λοιπόν ότι το 6-3-ε θα πρέπει να διαγραφεί, διότι έχουμε μία εσωτερική αγορά, δεν έχουμε τοπικές αγορές. Arvoisa puheenjohtaja, kollegat ja asiantuntijat, eh, on tärkeää, että turvallisuudesta. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κύριε Πυρογνώμονες, ε, είναι σημαντικό το ότι εδώ μιλάμε για την ασφάλεια προϊόντων και χαίρομαι που αναφέρονται και τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Αναφέρονται οι επικίνδυνες ουσίες. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε ε, στο μέλλον καταστροφές ε, όπως το θέμα του αμοιάντου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως και την αλλαγή του κλίματος όσον αφορά τα δομικά υλικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχους σχετικά με την ανάπτυξη και την αλλαγή του κλίματος. Στο παράρτημα 1 αναφέρονται τα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό όμως δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε ίσως στο άρθρο 6 τουλάχιστον ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι το carbon footprint, οι συνέπειες για το περιβάλλον. Έτσι να εξετάζουμε δηλαδή τις εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου κατά το σύνολο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίκο. Νομίζω ότι μίλησαν όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ως πρόεδρος και η συγκήτρια θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι προς τον κύριο Κούμανς. Μιλήσατε για ε, τους εργολάβους. Η ευθύνη ποιανού είναι κάτι που έχω μάθει από τον τομέα των ε, οικοδομών. Ε, είναι ότι πρέπει να κοιτάμε ποιο έχει την ευθύνη. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και δεύτερη ερώτηση. Ο κύριο Κούπερ ε, στην αρχή αναφέρθηκε στην καινοτομία. Ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτομία. Νομίζω ότι για πολλού ανθρώπου ε, που εργάζονται στον τομέα των οικοδομών. Ε, για πολλού ανθρώπου που εργάζονται στον τομέα των οικοδομών είναι χρήσιμο να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και το θέμα της γλώσσας είναι σημαντικό. Με ενδιαφέρουν λοιπόν δύο ερωτήσεις, το θέμα της ευθύνη ποιος είναι υπεύθυνο και το θέμα της καινοτομία. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο λοιπόν στους ομιλητές μας, παρακαλώ. Για το θέμα της ευθύνης, εν γέννη, αυτός που αναλαμβάνει το έργο φέρει την ευθύνη, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρξε κακοτεχνία, ελάττωμα στο προϊόν. Η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να αποδειχθεί αυτό εάν ο κατασκευαστής του προϊόντος δεν επιθυμεί να στηρίξει σε αυτήν την αιτίαση τον ε, ανάδοχο. Ο ανάδοχος τι είναι, μία μικρή εταιρεία. Ο κατασκευαστής κανονικά είναι μία πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί ε, ότι οφείλεται το λάθος ελαττωματικό προϊόν. Άρα την ευθύνη την πρωταρχική τη φέρει ο ανάδοχος, ε, ο εργολάβος ε, και άρα είναι, πολύ, είναι ζωτική σημασία να έχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το προϊόν. Ε, γιατί αν παραμείνει πελάτης επί σειρά ετών ο κατασκευαστής θα τον στηρίξει. Αν όμως ευκαιριακά αγόρασε κάτι από μια κατασκευαστική εταιρεία και έχει ένα γενικό πρόβλημα, γενικευμένο πρόβλημα με αυτό το προϊόν. Ε, ο κατασκευαστή ε, θα μετέλθει οποιοδήποτε νομικού μέσου κόλπου, μάλλον, για να ε, αποποιηθεί την ευθύνη. Μπορούμε να μείνουμε χρόνια εδώ και να το συζητάμε, αλλά να σας πω τι πιστεύω. νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιούμε απτά παραδείγματα ε, ε, κοιτάξτε αυτή την ράβδο ε, που χρησιμοποιείται σε μια δομική μέθοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε κάποιες άλλες χώρες αλλά όχι σε όλες για να συνδέσει δύο επιμέρους στοιχεία. Ε, μίας κατασκευής. Τέλος πάντων δεν είναι μόνο αγγλικό το προϊόν. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, γιατί ασχολείται με κάποια από τα ζητήματα του αποτυπώματος του άνθρακα, των επιπτώσεων δηλαδή του, στο περιβάλλον. Είναι πλαστικό, δεν είναι χαλίδινο ε, και έχει μεγαλύτερη επαγωγημότητα, δηλαδή χάνεται λιγότερη θερμότητα ε, έχει μικρότερη απαγωγημότητα και άρα χάνεται λιγότερη θερμότητα στους τοίχους. Ε, και το ε, τα πλαστικά προϊόντα δεν έχουν καλύτερη συμπεριφορά μέσα σε μια κατασκευή σε σχέση με τα χαλίδινα. Επίση είναι ενδιαφέρον γιατί ε, σκεφτείτε αυτό. Πώς θα το εξηγήσετε στους χρήστες. Αυτό έχει κέρια σημασία σε σχέση δηλαδή με το αν θα γίνει αποδεκτό ή όχι το προϊόν. Είναι σημαντικό οι αρχιτέκτονες που δεν είναι ειδικοί ε, να πάρουν κάποιε εξηγήσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος γιατί αλλιώς δεν θα το δεχτούν το προϊόν. Και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε το ETA, δηλαδή το περιεχόμενο και την ευελιξία ε, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή όλη, όλη η ενημέρωση που γίνεται στους ε, εργολάβους, στους αρχιτέκτονες ε, ε, πρέπει να είναι επαρκής ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά το προϊόν ο καθηγητής Μπόσε Μαΐρ μας μίλησε για ένα ευρωκώδικα. πώς το σχολιάζετε, ένα λεπτάκι να το σχολιάσω. οι ιδιότητες ε, των ε, προϊόντων όταν ε, θεωρούνται κομμάτι κάποιες κατασκευής κυρίως για παραδοσιακά προϊόντα ταξινομούνται σε κώδικες χρήσης. Το πρόβλημα με τα καινοτόμα προϊόντα είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιος κώδικας συχνά. Και άρα σκεφτείτε τις πληροφορίες που δίνετε στους χρήστες και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πώ ακριβώ θα παρουσιαστεί το προϊόν στους ε, χρήστε, Άρα δίκιο έχει ο καθηγητή. Από την... Αντίστροφα πρέπει να το πάρουμε. Αν υπήρχε κώδικας για όλα τότε και ήταν ε, λογικές οι πληροφορίες, ε, όλα θα ήταν τέλεια. Αλλά δεν μπορείτε βέβαια να έχετε όλα τα στοιχεία γιατί πάντοτε κάτι καινούριο θα κατασκευάζεται. Ο καθηγητή Μπόσεν Μαϊα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φοβάμαι πολύ την Κομισιόν. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον λόγο ευρωκώδικες. Θα ήθελα να μιλάω για τους ε, απλοποιημένους ε, ευρωπαϊκούς κανόνες ε, χρήσης. Και όσον αφορά το carbon footprint υπάρχει το TC350 για την αηφορία όπου υπάρχει ήδη για προϊόντα, και ελπίζω να τα λέω σωστά τώρα, PREN 15804 ε, που αναφέρεται σε όλα τα προϊόντα γενικά και έχει να κάνει με την περιβαλλοντική επισήμανση. Το carbon footprint, οι περιβαλλοντικές συνέπειες ε, του προϊόντος, αναφέρεται εκεί η ε, κατανάλωση ενέργειας που απαιτεί το προϊόν κλπ. Ελπίζουμε σύντομα, και αυτή είναι η ε, έκκληση υπαριθμών 7, ε, ελπίζουμε το 2013 να μπορούμε να έχουμε ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες, ε, να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση. Ξέρω ότι δεν μπορεί, η, δεν το Κοινοβούλιο να το επιφέρει αυτό εύκολα, αλλά ξέρω ότι έχετε τρόπους να το κάνετε και χρειαζόμαστε μάλλον και γι' αυτό το, το σημείο 7 ένα έγγραφο βάσης και θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριος Κούπερ. Στα βασικά αυτά έγγραφα θα πρέπει να αναφέρεται η έκκληση να, να υιοθετηθούν αυτά που ήδη έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, υπάρχει το θέμα του διαβατηρίου των κτηρίων. Όταν ε, έχουμε ευρωπαϊκούς εφαρμοστικούς κανόνες που εν μέρη αναφέρονται στην ε, ασφάλεια, την υγιεινή, το περιβάλλον, τη θερμομόνωση κλπ. Εάν κοιτάξουμε μαζί όλους αυτούς τους κανόνες, μπορεί για κάθε τέτοια παράμετρο να λάβουμε την πιστοποίηση που μας αξίζει, να το πω χοντρά. τελικά μπορεί να είναι τελείως παραπλανητικά τα πιστοποιητικά αυτά, κάτι που δεν θα γίνεται εάν έχουμε ένα πακέτο ευρωπαϊκών κανόνων. Το σημείο υπαριθμών 7 ταιριάζει πολύ καλά σε αυτό. Η αηφορία των κτηρίων σημαίνει οι εφαρμοστικοί κανόνες, δεν έχω τον αριθμό, αλλά ε, αυτό, μπορεί να μας το πει το, το CEN. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Μάγερ έθεσε μια ερώτηση, μην την ξεχνάτε παρακαλώ. Δεν ξέχασα καθόλου την ερώτηση του κύριου Μάγερ. Αυτό ακριβώς ε, θα επιχειρούσα να απαντήσω. Και χαίρομαι και για την ερώτηση που απευθύνεται στον κύριο Κούμανς. Και ευχαριστώ και τον κύριο Κούμανς για την ε, ειλικρινέστατη απάντηση που έδωσε. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα της ευθύνης και ποιος φέρει την ευθύνη για την εγκατάσταση ενός προϊόντος. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε πρώτα αυτό. Είναι θεμελιώδους σημασία. Για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας κύριε Μάγερ, αλλά είναι σημαντικό και για την αγορά. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο ότι έχουμε μόνο μία αγορά, την ενιαία αγορά, την εσωτερική αγορά και οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν έναν οδηγό για τη θέση των προϊόντων τους σε εμπόρια και αυτό το ρόλο παίζει ο κανονισμός. Ποιος όμως θα φέρει την ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων, μα οι εργολάβοι, μόνο οι εργολάβοι. Και χάρη στην ενημέρωση που θα έχουν, αυτοί θα αναλαμβάνουν την ευθύνη. Βέβαια υπάρχουν τόσες πιθανές χρήσεις και έχουμε και 27 χώρες μέλη. Κάθε χώρα μπορεί να έχει διαφορετικές απαιτήσεις για το κάθε προϊόν. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποτύχει ο κανονισμός σε ό,τι αφορά τις, δεσμεύσεις, τις υποχρεώσεις για κάθε προϊόν. Η αγορά είναι διαφορετική, όχι επειδή έχουμε 27 διαφορετικές χώρες μέλη, αλλά επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές πιθανές χρήσεις για ένα προϊόν. Και σε τελική ανάλυση την τελική ευθύνη τη φέρουν οι εργολάβοι. Οπότε αν δεν λάβουμε υπόψη αυτό το θέμα τη ευθύνη, ποιο είναι υπεύθυνο γιατί, και αν λάβουμε υπόψη και το γεγονό ότι υπάρχουν τόσε πολλέ ε, ε, δυνατότητες, εναλλακτικέ ε, ρυθμίσει εξαιτία τη εσωτερική αγορά και τη εφαρμογή αρχή επικουρικότητα, γιατί κάθε χώρα ρυθμίζει αυτό το θέμα και το, των χαρακτηριστικών. Είναι δύσκολο να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Την πολλαπλότητα των χρήσεων με την πολλαπλότητα των νομοθετικών διατάξεων. Γι' αυτό και δίνουμε στον εργολάβο που φέρει και τελική ευθύνη την δυνατότητα να επιλέξει το προϊόν και θα πρέπει να δώσουμε και στον κατασκευαστή μία ελαστικότητα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση που θα κάνουν προς τον εργολάβο. Αυτοί θα κρίνουν τι είναι απαραίτητο να γράψουν και για τη δική τους επιχείρηση. Γιατί στη Γερμανία, για παράδειγμα, η αγορά θα είναι πολύ αυστηρή. Και ο κόσμος, άσχετα με τη ρυθμιστική αρχή, θα είναι πολύ απαιτητικός για το προϊόν και πολύ πιο ακριβή στις ε, πληροφορίες που θέλει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα, για να μην πω λιγότερη αυστηρότητα. Βέβαια, μεγαλύτερη ελαστικότητα δεν σημαίνει και λιγότερη ασφάλεια υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή την ελαστικότητα στην αγορά, έχοντας υπόψη φυσικά ότι η τελική ευθύνη βαρύνει το χρήστη. Ο κύριος Μάγερ. Μία συμπληρωματική ερώτηση. Διότι στο άρθρο 6 σημείο 3 λέει ότι η, απόδοση, η δήλωση απόδοση θα πρέπει να περιέχει επιπλέον. Shall είναι υποχρεωτικό αυτό, δηλαδή δεν είναι προαιρετικό. Ο κατασκευαστής μπορεί να ε, αναφέρεται σε τοπικούς κανόνες, αλλά δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος να συμπεριλαμβάνει εκ των προτέρων ε, τους, ε, τις προδιαγραφές που ισχύουν σε κάθε μέρος της Ευρώπης. Εάν είναι προαιρετικό αυτό, εντάξει, αλλά όταν μιλάμε για ε, υποχρέωση, τότε δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον κατασκευαστή να ξέρει όλες τις τις τοπικές ιδιαιτερότητες στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα κλπ. Όχι υποχρεωτικά. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο, αλλά το άρθρο 3, και συμφωνώ απόλυτα, είναι του Συμβουλίου αυτό, παρόλο που το θέμα της, η έννοια της προτινόμενης χρήσης ε, θα πρέπει να συνδυαστεί με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Στα εναρμονισμένα πρότυπα, για παράδειγμα, που είναι εθελοντικά, γίνονται υποχρεωτικά αυτά αν υπάρχει ε, τοπική ρύθμιση ε, εθνική κάπου. Αυτό που αναφέρεται λέει ότι ο κατασκευαστής οφείλει, σαλ, οφείλει να δηλώσει την προτινόμενη χρήση ή προτινόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για όλους. Οι τεχνικές εναρμονισμένες προδιαγραφές είναι οι ίδιες για όλες τις χώρες είναι ακριβώς οι ίδιες. Ο κατασκευαστής πάντως είναι υποχρεωμένος να διαλέξει τουλάχιστον μία προτινόμενη χρήση. Και λογικά εφαρμόζεται το υπόλοιπο άρθρο. Αυτό δεν σχετίζεται με τις ε, αγορές, τις γεωγραφικές αγορές, δηλαδή την προέλευση ε, ενός προϊόντος. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια σωστή ενσωμάτωση του προϊόντος. Γιατί μερικά προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση το χειμώνα ή χρήση το καλοκαίρι. Άλλα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στην Ιταλία και άλλα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στι σκανδιναβικές χώρε. Θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αυτό. Και η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος επίσης είναι διαφορετική. Ε, ε, ή μερικά προϊόντα που έχουν συγκολητικές ικανότητες αν για τρεις μήνες μείνουν εκτεθειμένα στο ηλιακό φως χάνουν αυτή την ικανότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να φαίνονται. Να φαίνονται στο, στη σήμανση σε ε, ε, γιατί είναι διαφορετικές αυτές οι ιδιότητες για κάθε προϊόν. ανάλογα με το προϊόν και ανάλογα με τις ιδιότητες θα πρέπει να προσδιορίζονται οι χρήσεις. Για παράδειγμα, ορισμένα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην σκεπή είτε στο υπόγειο, αλλά δεν ισχύει αυτό για όλα. Θα πρέπει αυτό να φαίνεται ώστε αυτός που παραλαμβάνει το προϊόν στο εργοτάξιο να καταλαβαίνει αμέσως ε, για ποια χρήση προορίζεται. Θα ήθελα να πω ότι φυσικά έχει δίκιο ο καθηγητής Μάγερ με την ερώτησή του. Δεν μπορεί ένα προϊόν να πρέπει να επισημαίνεται ανάλογα με τον, τρόπο, με τον τόπο προορισμού του. Εμείς θεωρήσαμε αρχικά ότι ήταν λάθος στη μετάφραση, διότι στο, αγγλικό, στο γερμανικό κείμενο έλεγε όχι όπου τίθεται στην αγορά το προϊόν, έλεγε όταν τίθεται στην αγορά το προϊόν. Αυτό για νομικούς λόγους θα μπορούσε να το παραλείψει κανείς, διότι έχουμε ε, μια εσωτερική αγορά. Έτσι λοιπόν δεν έχει σημασία αν διατίθεται στην αγορά το προϊόν στη Μάλτα ή στο Βέλγιο. Το όπου όμως μπορεί να γίνει θέμα όταν τα κράτη-μέλη συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα, αυτό που είπε ο προλαλής σας, να επικαλούνται γεωγραφικές, ε, κλιματικές διαφορές, ιδιαιτερότητες, ώστε να ρυθμίζουν τα επίπεδα και τις κλάσεις. Αυτό διαφέρει από τις ε, τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Για... Όσον αφορά τον, ε, την προτινόμενη χρήση του προϊόντος δεν υπάρχουν ε, διαφορές εντός της Ευρώπης. Αλλά υπάρχει ένα τομέα όπου η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Το 63 ε λοιπόν διάταξη. Αντίκειται στην Ευρώπη. Ε, εάν έλεγα ότι θέλουμε να ε, πουλήσουμε προϊόντα στην Ελβετία, αλλά θα ήταν άδικο αυτό. Η Ελβετία είναι εκτός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στο αγγλικό κείμενο ε, αναφέρεται where, όπου ε, διορθώθηκε αυτό και γι' αυτό αντιδράμε. Διότι θα έπρεπε να λέει όταν τίθεται στην αγορά. Εάν πω όταν, δεν χρειάζομαι κανέναν ορισμό της εσωτερική αγοράς και απλά μπορώ να διαγράψω τη φράση αυτή. Αυτό απλοποιεί κάπως τον κανονισμό. Ο κύριος Φερτάιζεν είναι εδώ ακόμη. Θέλει να σχολιάσει πάλι αυτό το θέμα ή θέλει να κάνει μια επερώτηση ίσως. Ε, μάλιστα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Je vais Θα ήθελα μόνο να διευκρινίσω το εξής. Αυτό που προβλέπετε εδώ, στα γαλλικά, στο 6-3-ε, έτσι, 6-3-ε, όχι α, ε. ε la référence qui Η αναφορά λοιπόν που γίνεται εκεί είναι ε, ο τόπος όπου τίθεται σε εμπορία το προϊόν. Δηλαδή, ο κατασκευαστής θα ξέρει εξ ορισμού πού θα διαθέσει, σε ποια αγορά θα διαθέσει το προϊόν του. Η πρώτη εμπορική συναλλαγή ισοδυναμεί με τη θέση σε εμπορία. Άρα, άρα υπάρχει θέση σε εμπορία με το που ε, πουλήσει το προϊόν ο κατασκευαστής και άρα θα πρέπει να υπάρχει γνώση των εθνικών απαιτήσεων για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ε, από ό,τι κατάλαβα φοβάστε ότι είναι ευρύτερη διάταξη, αλλά δεν είναι. Μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά μιλάμε για ένα συγκεκριμένο τόπο. Μπορεί να είναι γερμανική κατασκευαστική εταιρεία που ε, θέτει σε εμπορία στην Ιταλία ή στη Γαλλία ένα προϊόν, αλλά εκεί θα θεωρηθεί ότι εισέρχεται στην ε, ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Αυτά τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένη χώρας πρέπει να λάβει υπόψη. Δεν νομίζω ότι θα ε, έπρεπε να ανησυχούν γι' αυτό οι κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά μπορεί να έχω και άδικο. Ε, <laughs> Η Επιτροπή ζητώ συγγνώμη. Ε, γιατί ε, άκουγα για το 3-6α ενώ μιλάμε για το 63 3 εδώ πέρα γι' αυτό καμία σχέση με την απάντηση που σας έδωσα προηγουμένως ε, τώρα καταλαβαίνω και καλύτερα το ερώτημά σας πολύ δυσεπίλητο αυτό το θέμα I think that's coming to the end of our Τώρα πλησιάζουμε στο τέλος της ακρόασής μας. Θα ήθελα να συνοψίσω εντάχει. Τροφοδοτήσατε σε μεγάλο βαθμό τον προβληματισμό μας. Ήταν εξαιρετικοί οι επιστημονικοί συνεργάτες που καλέσαμε. Ε, το θέμα της ε, χρηματοδότησης ε, των ETAs, των DDAs, e για, ε, τον κατασκευαστικό κλάδο και τα δομικά υλικά και τις ιατικές εξαιρέσεις σίγουρα θα ξανασυζητηθούν πολλά και σε αυτά τα θέματα. Ε, κάτι που συγκράτησα είναι το θέμα της αστυνόμευσης για τη σήμανση ΕΚ. Ε, με περικοπές στον προπολογισμό, τα κράτη-μέλη δεν ξέρω πόσα ακριβώς θα έχουν επαρκείς πόρους για να επιβλέψουν ε, την εφαρμογή για να υπάρχει ασφάλεια και να διατηρηθεί η ποιότητα των των προϊόντων, τι πρέπει να δηλωθεί τώρα, αν πρέπει να δηλωθούν οι επικίνδυνες ουσίες ή όχι, η χρηματοδότηση των αρχών, η ευθύνη του κατασκευαστή και του εργολάβου, το θέμα των μικροεπιχειρήσεων. Ε, όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία θα μας προβληματίσουν εδώ στην Επιτροπή στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ ε, τα μέλη που έμειναν μέχρι τις 6 παρα 10. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους ε, των βουλευτών, των βιομηχανικών κλάδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ακρόαση.